Uh, Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους έφτασαν μόλις τώρα και για όσους ε, ήταν εδώ από το πρωί, σας καλημερίζω ξανά. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού αποφάσισε να οργανώσει αυτή την ακρόαση με τους γενικούς διευθυντές από ορισμένες γενικές διευθύνσεις για να δώσει τη δυνατότητα στη διοίκηση να ενημερώσει τα μέλη για την ε, δομή της υφιστάμενης εργασίας και για τα σχέδια που δρομολογούνται για το 2021 εν ώψη της σύνταξης της έκθεσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού από πλευράς αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Σας καλωσορίζω όλους. Θέλω να σας παρακαλέσω να τηρήσουμε αυστηρά το πρόγραμμα να εκτελέσουμε τη χορογραφία ακριβώς όπως πρέπει ή αλλιώ θα ξεπεράσουμε το χρονικό όριο που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Ε, θα δώσω στον ε, κύριο Πετή 10 λεπτά για την έκθεσή του και θα δώσω 5 λεπτά στις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις και πραγματικά θα διακόψω αυτόν που θα ξεπεράσει το χρονικό διάστημα που του έχω παραχωρήσει. Να τηρήσουμε παρακαλώ αυστηρά το χρονοδιάγραμμα και στη συνέχεια τα μέλη που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις μπορούν να τις θέσουν για ένα ολόκληρο λεπτό, όχι παραπάνω. Παρακαλώ να θέτετε ερωτήσεις ακριβείς, συγκεκριμένες, για να μπορούν και οι αρμόδιοι από τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις να είναι σε θέση να απαντήσουν. Ξεκινούμε λοιπόν ευθύ αμέσω. Καλωσορίζω τον κύριο Πλατή, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει να προσκαλέσετε διάφορες γενικές διευθύνσεις, διάφορες εκπροσώπους αυτών για την οικονομική χρήση 2021 και για τις ε, ε, δραστηριότητες που απορρέουν από αυτή. Πέρα από την ε, ονοματολογία και τον όγκο, εγώ και οι συνάδελφοι θέλουμε να σας παρουσιάσουμε πώς ε, αντιλαμβανόμαστε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποια είναι, ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Σκοπός είναι να βοηθηθεί ο βουλευτής για τις, να ασκήσει τις του δραστηριότητες. Μιλώ ως διοικητικός αρμόδιος υπεύθυνο για την σύνταξη του προϋπολογισμού και Είμαι υπεύθυνο επίσης και για, ε, ε, ε, και για τα οικονομικά των βουλευτών και των βουλευτικών γραφείων. Θα σας υπενθυμίσω δηλαδή τη διοικητική και οικονομική διαδικασία η οποία μας, δεί, μας δείχνει πόσο υιοθετείται προσωρινά το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε ποιες κατευθυντήριες ε, γραμμές κινείται και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις ειδικέ πιστώσεις της Γενικής Διεύθυνσης για τα οικονομικά. Ε, σύντομη, να σας παρουσιάσω ποιοι είναι οι τομείς δραστηριότητας της DG Fins και κάποια βασικά αριθμητικά στοιχεία που δείχνουν τη δραστηριότητά της. Η DG Fins έχει λοιπόν τρεις ε, διευθύνσεις, 282 ε, υπαλλήλου. 20% είναι συμβασιούχοι και το υπόλοιπο είναι μόνιμοι. 60% υπηρεσίες είναι στις Βρυξέλλες και 40% στο Λουξεμβούργο. Συνολικός προϋπολογισμός είναι 426 εκατομμύρια για το 2021. Η διεύθυνση Α, Budget και Financial Services, τέσσερις μονάδες, κάνει το συντονισμό των εγκάρσιο και στηρίζει τις άλλες υπηρεσίες του ε, Κοινοβουλίου. Η μονάδα για το budget, για τον προπολογισμό, κάνει το συντονισμό του προπολογισμού των διαφόρων υπηρεσιών. Έχουμε την κεντρική οικονομική μονάδα που βοηθά για τα κανονιστικά και νομοθετικά θέματα. Έχουμε το τη διεύση για τα λογιστικά, όπου εκεί διασφαλίζονται αποκλειστικά τα θέματα του Ταμείου και της διαχείρισης των ροών. Και έχουμε και τμήμα για την πληροφορική με βάση το FMS, ορισμένα σημαντικά αριθμητικά στοιχεία. Ύψος πληρωμών 1 δις 840 περίπου εκατομμύρια το 2019. 658 εκατομμύρια συναλλαγές, 26 εκατομμύρια τιμολόγια, μεταξύ άλλων. Ε, υπάρχει διαδικτυακή πύλη των μελών είναι το σημείο επαφής μεταξύ των βοηθών για να υποβάλλονται εκεί τα αιτήματα επιστροφής ε, χρημάτων και να έχει κανείς ενημέρωση για τα έξοδα που καλύπτονται και τρεις ειδικέ μονάδες για το μισθολόγιο, για τα εργασιακά, για την κοινοβουλευτική βοήθεια και για την επιστροφή των εξόδων μετάβασης και ε, διαβίωσης. 234 εκατομμύρια ευρώ διαχειρίστηκε. Ε, πάρα πολλές αιτήσει είναι αυτές που υποβάλαμε. 8.268 συμβάσεις έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας. 218.000 ε, συναλλαγές για την εκαθάριση των εξόδων ταξιδίων. Βλέπετε τεράστιο όγκο συναλλαγών. Τέλος, η Διεύθυνση ΣΥ ασχολείται με τη χρηματοδότηση των πολιτικών δομών και τη διαχείριση των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Έχουμε βασική χρηματοδότηση των πολιτικών ομάδων και των πολιτικών ιδρυμάτων, βοήθεια για τους μη εγγεγραμμένους, βλέπετε τα αντίστοιχα νούμερα. Δεύτερο μέρος της παρουσίασής μου πολιτική και διοικητική διαδικασία για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2021. Είναι μια διαδικασία που εκτείνεται σε διάφορους μήνες και έχουμε τις προτεραιότητες και τα ύψη των πιστώσεων τα οποία καταρτίζονται. Γίνεται διοικητικό σχέδιο το οποίο υποβάλλεται σε διαιτησία από εμάς, από εσάς και τελική απόφαση. Βλέπετε στη διαφάνεια τη διαδικασία η οποία γίνεται για 4-5 μήνες. Έχουμε τη διοικητική φάση και την πολιτική φάση. Για την πολιτική φάση είστε εσεί υπεύθυνοι. Ποια είναι η παραδοσιακή αλληλουχία των γεγονότων. Έχουμε μια προπαρασκευαστική φάση. Ε, δίνεται ένα σημείωμα στους εντολείς να αναλύσουν τις αιτήσει και γίνεται ακρόαση με τις γενικές διευθύνσεις. Στη συνέχεια έχουμε διατησία με το Γενικό Γραμματέα και οριστικοποίηση της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για το προσχέδιο για τις προβλέψεις, αυτό που σας παρουσιάστηκε χθες. Χθες λοιπόν ξεκίνησε η πολιτική φάση με την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και στη συνέχεια έχουμε φάση συνδιαλλαγής. Το προσχέδιο από το Προεδρείο, το αντίστοιχο της Επιτροπής σας και το αντίστοιχο στην Ολομέλεια στη συνέχεια. Σε αυτή τη διαδικασία θέλω να σταθώ σε δύο σημεία που δεν γνωρίζετε πολύ καλά τα αποτελέσματα της ακρόασης και τις εντολές στους, ε, που δίδονται στους εντολείς. Όταν προετοιμάζουμε αυτό το αίτημα για το προϋπολογισμό, καλούμαστε να επιδιώξουμε κοινού στόχους που απορρέουν από τις πιο πρόσφατες πολιτικές επιδιώξεις, με βάση τις αποφάσεις του Προεδρείου που απορρέουν από τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, όπως προβλέπεται από τον οικονομικό κανονισμό. Στους στόχους του 2021 θέλω να υπογραμμίσω αυτά που τόνισε και ο συγητής χθε, δηλαδή ότι η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαρτάται από την ικανότητά του να διαχειριστεί σωστά τις δικές του δαπάνες με βάση τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μπορεί να εγκρίνει και τους προϋπολογισμούς των άλλων θεσμικών οργάνων. Έχουμε 200 γραμμές στο προϋπολογισμό και κάθε ένας από τους εντολείς ε, εξετάζει κάθε μία από τις γραμμές, ποια σχέδια δρομολογήθηκαν, ποια ολοκληρώθηκαν, ποιες είναι οι νέες δραστηριότητες με και αριθμητική ε, αναπαράσταση με νούμερα δηλαδή αντίστοιχα και στο, έχουμε την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου, την αποχώρηση και ε, τις νέες προτεραιότητες του πολιετούς δομεσονομικού πλαισίου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά για τη χρήση του 2021. Τα αποτελέσματα ε, των ακροάσεων δίνουν ε, ενδιαφέροντα συμπεράσματα έγινε μια πρώτη ανάλυση των ετοιμάτων των γενικών διευθύνσεων και ορίσαμε τις ανάγκες της κάθε γενικής διεύθυνσης στο έπακρον και τις ανάγκες τους για αύξηση ή μείωση των επιστώσεων. Έχουμε 1,6% αύξηση σε σχέση με τα αρχικά αιτήματα των εντολέων. Και θα γίνει μια πρώτη διαιτησία με το Γενικό Γραμματέα γιατί βλέπετε ότι υπάρχει απόκληση στα νούμερα. Τώρα περνάω στο τρίτο μέρος της παρουσίασής μου, τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τη χρήση 2021. Θα παρουσιάσω τις παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε, τις προτεραιότητες της οικονομικής χρήσης 2021, ε, τη μεγάλη δημοσιονομική μάζα, δηλαδή προς τα που στρέφεται ο κύριος όγκος του προϋπολογισμού, το πώς κατανέμονται οι υποχρεωτικές δαπάνες και οι προσαρμόσιμες δαπάνες, ε, τις δαπάνες για την πολυγλωσία και ούτω καθεξής. Ποιες είναι οι παράμετροι. Οι παράμετροι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την αξιολόγηση των πιστώσεων. Θέλουμε να εναρμονίσουμε την προετοιμασία των εντολέων και να εναρμονίσουμε το εγχείρημα μας με αυτό των άλλων θεσμικών οργάνων. Και επίσης το ποσοστό του πληθωρισμού που περιμένουμε ανάλογα με τα είδη των δαπανών με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν στο καταστατικό για τις δαπάνες. Δεν αναπαράγουμε τις πιστώσεις από τη μία χρόνια στην άλλη, δεν κάνουμε απλά copy-paste, αξιολόγουμε κάθε φορά κατά πόσο αυτές είναι αναγκαίες και κατά πόσο ανταποκρίνονται ε, στον τιμάριθμο και στην εξέλιξη των τιμών. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε χθε τις προτεραιότητες για την οικονομική χρήση 2021, οι οποίε είναι οι εξή. η επικοινωνία με τους πολίτες, το κτηριακό πρόγραμμα που εκτείνεται σε πολιετή βάση, ε, ένα ε, εξυγχρονισμό των υποδομών ε, των υποδομών διασκέψεων, την ασφάλεια, την πληροφορική και το πρασίνισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Κτηρίων, μεταξύ άλλων. Βλέπετε εδώ πώς ε, κατανέμεται ο κύριος όγκος του προϋπολογισμού. 712 εκατομμύρια ευρώ, 34% των πιστώσεων. Είναι η πιο μεγάλη δαπάνη για τους μονίμους, για το μόνιμο προσωπικό. Μετά έχουμε τις άμεσες δαπάνες των βουλευτών, 431 εκατομμύρια, 20% πιστώσεων. Τρίτο σημαντικό ε, στοιχείο είναι οι δαπάνες για τα κτίρια και τις υποδομές, 253 εκατομμύρια, 12% του συνόλου των πιστώσεων. Άρα 66% του προϋπολογισμού έχει να κάνει με το προσωπικό τους μονίμως τους βουλευτές και το κτίριο και τα κτηριακά. Το 34% που μένει πηγαίνει στην πολυγλωσία, στην πληροφορική, στις εκστρατείες επικοινωνίας και στις δαπάνες των πολιτικών ομάδων. Σε αυτή τη διαφάνεια τώρα βλέπετε πώς κατανέμεται ο προϋπολογισμός μεταξύ δαπανών οι οποίες εντάσσονται σε υποχρεώσεις του καταστατικού και δαπάνες που απορροκύπτουν βάσει συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός για να αξιολογήσουμε αν έχουμε περιθώριο λιγμών στο πώς θα χειριστούμε τις πιστώσεις. Στην πρώτη κατηγορία δεν υπάρχει ευελιξία, ούτε σε όγκο ούτε σε εξέλιξη τιμών. Έχουμε εξέλιξη των τιμών σε σχέση με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ο αριθμός των μονίμων ε, ορίζεται από το οργανόγραμμα και η εξέλιξη των μισθών ακολουθεί την ίδια μέθοδο με αυτήν ε, που ακολουθείται για τους μισθούς των βουλευτών. Τώρα, στις διοικητικέ δαπάνες που προκύπτουν ε, από συμβάσεις, οι κανόνες για την τιμαριθμοποίηση στις συμβάσεις έχουν να κάνουν με τον όγκο των δαπανών. Άρα, το αληθινό περιθώριο λιγμών έγκυται στις επενδύσεις. Και όντως αυτός ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει αντικείμενο διατησίας. Συχνά τίθεται ερωτήματα για το κόστος της πολλαγλωσίας που είναι μοναδικό, ε, μοναδική διαμορφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. 459 εκατομμύρια συνολικά, 22% του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Έχουμε τις άμεσες και έμεσες δαπάνες, 428 εκατομμύρια οι δαπάνες του προσωπικού και τα υπόλοιπα οι έμεσες. Οι συνάδελφοι, οι γενικοί διευθυντές θα παρουσιάσουν το προϋπολογισμό τους ο καθένας. Εδώ βλέπετε πώς κατανέμε το προϋπολογισμό μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Οι πιο μεγάλες δαπάνες δεν μας εκπλήσει ότι είναι στη Γενική Διεύθυνση για το προσωπικό. 1 δις 34 εκατομμύρια, τη Γενική Διεύθυνση ΦΙΝΣ με 426 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές. Θα ολοκληρώσω εστιάζοντας την προσοχή μου στις πιστώσεις της DG Finance. Δαπάνε σε σχέση με τους βουλευτές. Η βοηθή. 215 εκατομμύρια για την οικονομική χρήση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δαπάνη. Τα άλλα είναι περίπου αντίστοιχα σε όγκο, δηλαδή η μισθή των βουλευτών, και τα έξοδα ταξιδίου μετάβασης περίπου είναι το ίδιο. Γενικές δαπάνες ε, αντιστοιχούν σε 40 εκατομμύρια περίπου. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη διαφάνεια γιατί μας δίνει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα που τέθηκαν χθε. Αξιολόγηση της βοήθειας των βοηθών γίνεται με θεωρητικό τρόπο. Αριθμός των βουλευτών επί χ εκατομμύρια ευρώ επί 12 μήνες και σε σχέση με την ιστορική χρήση που έχουμε διαπιστώσει οι βουλευτές ε, αξιοποιούν περισσότερο το χρηματοοικονομικό τους φάκελο και όλο και περισσότερο ε, προσλαμβάνουν τέταρτο βοηθό και ε, ασκούμενο με αμοιβή. Και έτσι αυξάνονται τα ποσά παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των βουλευτών είναι μειωμένος. Ήταν ήδη μειωμένος για τη χρήση 2020 γιατί τον Ιανουάριο έχουμε τους 751 μέση τιμή του ταξιδιού που έχουμε παρατηρήσει. Με βάση αυτή υπολογίζουμε ε, τις δαπάνες ταξιδίου σε σχέση με το παρουσιολόγιο των βουλευτών και ε, την κίνηση. Αυξάνονται λοιπόν τα έξοδα ταξιδίου στις, ε, όταν έχουμε μείνει σύνοδο στις Βρυξέλλες και αυξημένες δαπάνες, 900.000 παραπάνω το χρόνο. Αυξάνονται οι δαπάνες για το Στρασβούργο, και έχουμε και πληθωρισμό 2,3% για αυτά. Τέλος. Εδώ το κόστος της χρηματοδότησης των πολιτικών δομών, προσωπικό των πολιτικών ομάδων, περίπου 112 εκατομμύρια ευρώ. Δαπάνες για τη λειτουργία των πολιτικών ομάδων 65 εκατομμύρια, 46 εκατομμύρια χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και χρηματοδότηση πολιτικών ιδρυμάτων ευρωπαϊκών 23 εκατομμύρια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε πέντε λεπτά χρόνο παραπάνω θα σας ε, το δώσω γιατί είναι σημαντικό, αλλά για τις υπόλοιπες γαμαδέλτα πέντε λεπτά γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Να δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές να θέσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Σαστέλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικά Διευθυντά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Την απαντήστε την πρώτη γιατί την έθεσα και στο Γενικό Γραμματέα χτες. Είχε να κάνει με την αύξηση του κονδυλίου για τη βοήθεια των βουλευτών. Την απαντήσατε όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι δαπάνες ταξιδίου. Απαντήσατε και σε αυτό δεν σας δω περαιτέρω εξηγήσει. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει όχι τόσο με τις εργασίες για το αντενάουερ, για το κτίριο αντενάουερ αλλά για τον τρόπο χρηματοδότησης. Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του Ραμασάζ και φαίνεται να μας λέτε ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε και για τη νέα πτέρυγα, τη δυτική, και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική του Ραμασάζ σε σχέση με τον οικονομικό αντίκτυπο και το κόστος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, ο τρόπο χρηματοδότηση είναι στα χέρια σα. Εμεί. έχουμε παρουσιάσει πριν από ε, κάθε σχέδιο για τα κινήτα και για τα κτίρια στο Λουξεμβούργο. Προσφύγαμε στην Επιτροπή προπολογισμών όταν επρόκειτο να υιοθετηθούν ε, αυτά τα σχέδια. Όταν υιοθετείτε το σχέδιο έχετε την χρηματοδότηση στο πλαίσιο των 450 εκατομμυρίων που μπορεί να γίνει είτε προσφεύγοντα σε δάνειο τώρα είναι δυνατόν ε, με τον θεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό εδώ και δύο χρόνια ή γράφοντας τις ανάγκες χρηματοδότησης ε, για το δάνειο που ε, χρειάζεται στον προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη χρονιά. Όμως ε, υπάρχει ουσιαστικά απόκληση της χρήσης από το ένα έτος στο άλλο γιατί οι πιστώσεις χρηματοδότησης δεν αφαιρούνται από τις διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, τις κανονικές αν η Δημοσιονομική Αρχή αποφασίσει να δώσει επιπλέον 100 εκατομμύρια τη χρονιά και είναι απαραίτητα αυτά τα εκατομμύρια για την κατασκευή. Μπορούμε να το έχουμε στη γραμμή του προπολογισμού. Όμως, αν δεν περάσει στη γραμμή του προπολογισμού, αν έχουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στον προπολογισμό, μπορεί να έχουμε 2 ή 3% των πιστώσεων που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί. Είμαστε πολιτικό οίκο, κάποια πράγματα γίνονται ή δεν γίνεται. Περνούν χάρη, μπορεί να καθυστερήσουν οι διαγωνισμοί για του υπολογιστέ. Ε, ε, η αρχή ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε έλλειμμα στο τέλος του έτους. Χρειάζεται λοιπόν ένα ε, ποσοστό 1% θα έλεγα, ένα περιθώριο ασφάλειας. Η δυνατότητα υπάρχει στο τέλος του έτους να ενεργοποιηθούν αυτά τα ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και μόνο η Δημοσιονομική Αρχή μέσω ουσιαστικά εμβάσματος πιστώσεων αποφασίζει αν θα το κάνει ή όχι. Και η δυνατότητα είναι ότι κατά τη διάρκεια της ε, κατασκευής ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ποσά που έχουν ενεργοποιηθεί και για να αποφύγουμε τους ε, μετέπειτα τόκους που συσσωρεύονται από τη στιγμή που ολοκληρώνεται ένα έργο και τη στιγμή της αποζημίωσης του δανείου που θα πρέπει να γίνει στο τέλος και τους διάφορους τόκους από το δάνειο που θα προέκυπταν. Έτσι λοιπόν, ε, τέλος πάντων αυτά ποσά πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούν ε, και το να τα πληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για τα επόμενα έτη και σας δίνει περισσότερη δυνατότητα για επιλογές ε, γιατί δεν θα έχουμε αυτό το άχθος τα επόμενα έτη για την ε, δική μας δίκηση λοιπόν όταν το εγγράφουμε είτε το εγγράφουμε στην αρχή ε, του οικονομικού έτους είτε γίνεται ενεργοποίηση στο τέλος υπάρχει διαφορά για μας όμως νομίζω ότι είναι καλό να διατηρηθεί η ευελιξία για το έτος και να μην πληρώνουμε ε, το κους ούτε για τα δάνεια ούτε μετέπειτα το είναι νομίζω καλό να ενεργοποιούνται και οι δύο τρόποι για τις πιστώσεις που έχουν απομείνει στο τέλος του έτους. Κύριο Σούζεκοφ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση αφορά το Brexit. Είναι δυνατόν να έχουμε όλες τις πληροφορίες για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού για το πώς ε, πλήττει τον προϋπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκονομήσουμε χρήματα. Γιατί φεύγουν ε, οι συνάδελφοι από την Βρετανία και φαίνεται ότι εμείς ε, θα δαπανίσουμε περισσότερα. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να έχουμε ένα πίνακα και δεύτερη ερώτηση για τη μεθοδολογία. Προσπαθώ να καταλάβω αν ε, έχουμε αποτελέσματα τα χρήματα που δαπανώνται. μα είπαν χτες ότι 8,06% αύξηση στην συμμετοχή σε εξηγείται από τις αυξημένες δαπάνες ε, στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι εξηγείται αυτό, ε, όμως ε, αυτό πράγματι έχει οδηγήσει στην αυξημένη συμμετοχή. Πώς εκτιμούμε ότι το 8% συνδέεται με τις δαπάνες του Κοινοβουλίου. Και άλλη φορά μας είπαν ότι αυξάνονται οι επισκέπτες στον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ε, μπορούμε να μας δώσετε κάποια κάποια ένδειξη για τα αποτελέσματα που έχουμε. Θα ήθελα να δω λοιπόν ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ νομίζω είναι αρμόδια για το τελευταίο τμήμα τη ερώτησή σα. Να απαντήσει τώρα ο κ. Κλητή για, την υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των Βρετανών συναδέλφων σας. Καταρχήν είχαν εγγραφεί στον προπολογισμό του 2020 γιατί είχαμε πιστώσει μόνο για τον Ιανουάριο και όχι για τους επόμενους μήνες τώρα. Σε ό,τι αφορά τις εξοικονομήσεις, όλες ε, οι θέσεις δεν ε, ε, εξαφανίστηκαν γιατί από 751 πάμε στους 705 βουλευτές γιατί Έχουμε 27 έδρες που αναδιαναμήθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν έχετε εξοικονομήσει 46 θέσεων. Ένας βουλευτής κατά μέσο όρο κοστίζει 500 ε, έως 600 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε έναν αριθμό γραμμών του προπολογισμού ε, που μειώνονται, όμως ε, το, στο 21 έχουμε και τις μεταβατικές αποζημιώσεις για τους Βρετανούς βουλευτές, δηλαδή ε, όσοι ήταν εδώ για πολύ καιρό θα λάβουν αποζημίωση για 24 μήνες, την αποζημίωση για το μισθό σας. Έτσι λοιπόν, να πω ότι το 46 είναι μικρός αριθμός ε, για να μπορεί να ε, έχει αντίκτυπο. Δεν ε, μπορούμε, παίρνουμε το χάρη, να καταργήσουμε 16 γραφεία. Όμως, επειδή θα έχουμε δύο-τρεις βουλευτές Βρετανούς λιγότερους, δεν θα δούμε πραγματική μείωση στο κόστος. Το άμεσο κόστος των βουλευτών που φεύγουν μα ενδιαφέρει και έχουμε υπολογίσει όλε τι γραμμέ προπολογισμού σε σχέση με τι άμεσε δαπάνε των βουλευτών με 500 βουλευτέ για το 2021 και όχι για 751. Λοιπόν, για την εκλογική εκστρατεία θα αφήσω τη συνάδελφο από την ΓΑΜΑ να απαντήσει τώρα για τις πολιτικές ομάδες και τα κόμματα. Οι πολιτικές ομάδες δεν είχαν πρόσθετες πιστώσεις ε, για την προεκλογική εκστρατεία, όμως ε, τα κόμματα και τα ιδρύματα είχαν λάβει πιο αυξημένα ποσά, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό 1141 που προσδιορίζει τη γνωτήση των κομμάτων και των ιδρυμάτων, ε, έχουν τα κόμματα ένα ρόλο διάρθρωσης της πολιτικής σκέψης στην Ευρώπη. Και ε, ουσιαστικά είναι αρμόδια για να διαδώσουν ε, τα κύρια ρεύματα ιδεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν τα ευρωπαϊκά κόμματα έλαβαν τα κονδύλια σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα. Δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός ε, που έχουμε στην αντίστοιχη γραμμή προϋπολογισμού κατανέμεται σύμφωνα με τον αριθμό των βουλευτών που είναι μέλη του κάθε Ευρωπαϊκού Κόμματος. Κύριε Αρμό. I just want to, to, uh... Ε, θέλω να ομολογήσω και ζητώ συγγνώμη που κατέθασα λίγο καθυστερημένη, αλλά τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, συγκρίνουμε τον ε, προπολογισμό για το 2021 με αυτόν του 2020 ή με την πραγματική δαπάνη που έχει λάβει η χώρα στο παρελθόν και πώς ακριβώς το κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Ευχαριστώ έχουμε πάντοτε ένα ενδιαφέρον δείκτη, να έχουμε ε, το ποσοστό αύξηση από το ένα έτος στο άλλο. Γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας σας μίλησε για το ποσοστό του 3,2%. Τι ε, συμβαίνει εδώ, όπως εξεκριμένο. Ξεκινάμε από έναν όγκο δραστηριοτήτων ε, που εκτιμούμε και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη των τιμών ε, που ισχύουν για αυτό τον όγκο δραστηριοτήτων για τους μισθού των μολύμων παραδείγματος χάρη και των βουλευτών. Έχουμε τη αριθμητική αναπροσαρμογή που προβλέπεται στον κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που είναι η μέθοδος για τους μισθού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, μιλάει ε, για 2,6% ε, και ε, μετά έχουμε 2,5% από τον Ιούλιο του 2020 και αυτό εφαρμόζεται για την εκτίμηση των μισθών των βουλευτών και του μονίμου προσωπικού. Για άλλες αποζημιώσεις γενικών δαπανών ή για τις αποζημιώσεις για τα ταξίδια και τη διαμονή έχουμε ε, τον ε, τιμάριθμο της 1ης Οκτωβρίου κάθε έτος που ισχύει και υπάρχει εναρμονημένη εναρμόνιση της Κομισιόν που εφαρμόζεται στο σύνολο του προπολογισμού. Και έχουμε μια τρίτη κατηγορία που είναι οι συμβάσει. Εδώ εφαρμόζουμε την ρήτρα που προβλέπεται στις συμβάσεις για την παιχνιδική προσαρμογή, εκεί όπου εκτελούνται οι συμβάσεις. Αν μιλάμε για πρόσληψη στο Λουξεμβούργο, σίγουρα θα ισχύσει ε, το ότι ισχύει για το Λουξεμβούργο, για μια σύμβαση στο Παρίσι. Ε, Παραδείγματο χάρη θα έχουμε τον ε, την εθνική προσαρμογή που αντιστοιχεί στο Παρίσι και τα κτλ. Έτσι λοιπόν σε κάθε κατηγορία δαπανών ε, εφαρμόζουμε ε, το συντελεστή ε, που αφορά την αύξηση των δαπανών και αυτό μπορεί να αφορά αύξηση των δαπανών από το ένα έτος στον άλλον και ουσιαστικά εκεί βλέπουμε τις διαφοροποίησεις μεταξύ του συνόλου του προϋπολογισμού του 2020 2021. Ο κ. Ναι, ένα-δυο παρόμοια ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Ε, καταρχήν, ε, αυτές οι γραμμές οι οποίες σχετίζονται ε, με τις ε, δαπάνες των ευρωβουλευτών αυξάνονται και εκείνες, στην πρικοδότηση δηλαδή. Αν έχουμε πραγματικά λάβει υπόψη μας τις επιπτώσεις του Brexit, τότε θα πρέπει να το δούμε και αυτό στις γραμμές να πηγαίνει. Γιατί αν δούμε για παράδειγμα τις ταξιδιωτικές δαπάνες και για τους ευρωβουλευτές αλλά και για το μόνο προσωπικό, αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες, και για παράδειγμα από τη Γραμματεία και από τις ε, πολιτικές ομάδες. Σε όλες αυτές ε, λοιπόν τις γραμμές ε, θέλαμε, ελπίζαμε να δούμε μία μείωση αλλά βλέπουμε αύξηση οπότε θα θέλαμε να, να μας εξηγήσετε λίγο από πού έρχονται αυτές τις αυξήσεις. Ποιο, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή, αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Μετά σε ό,τι αφορά το, αυτό το greening όπως λέμε του υπροπολογισμού. Ε, νομίζω πως δεν αναφέρονται πολλά σε ό,τι αφορά τι επιπτωσει ε, ε, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες διοξιδίου του άνθρακα, σε ό,τι αφορά τι επιμέρους γραμμές και νομίζω πως αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα κτίρια, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά αυτή την αύξηση τη της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2,3% και το πώ έχει επίπτωση στις ε, ακριβώ στι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, από πού έχει προέλθει αυτό. Ε, θα πρέπει να καταστήσουμε πιο βιώσιμο τον προπολογισμό σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτέ τι εκπομπέ. Ευχαριστώ. Ε, βέβαια, το τελευταίο σχόλιο που κάνατε αφορά την ηλιο ε, και όχι τον κύριο Κλέντο. Οπότε ο κύριο Κλέντο για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ. Και πάλι αν συγκρίνουμε τον προπολογισμό του 2021 με το 2020, σε ό,τι αφορά και βάσει των αριθμών των βουλευτών θα πρέπει να έχουμε κατά νου του 20 είχε υπολογιστεί 11 με 11 μήνες και ε, είχαμε εκεί τους περισσότερους βουλευτέ και ε, έτσι λοιπόν είχαμε ένα πρόσθετο προπολογισμό που συμπληρώθηκε για τον Ιανουάριο του 2020. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη στον όγκο των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων ε, το απαντήσατε αυτό, κύριε Κλετή. Η ίδια ερώτηση τέθηκε και είναι η ίδια η απάντηση. Επόμενο μιλήτρια. Uh, Σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε ε, Ναι, αναφερθήκατε στους ευρωβουλευτές, αλλά έχουμε και 150 λιγότερους βοηθούς. Ε, αυτό δεν έχει επίπτωση στον προπολογισμό. υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία θα πρέπει να εκταμιευθούν ακόμα. I think that has already been answered. Uh, Κύριος ε, ε, νομίζω πως αυτό απαντήθηκε προηγουμένως κατά την αρχική παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Κλέτη. Κύριε Κλέτη, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, κύριε Κλέτη. Οι βοηθοί δεν πληρώνονται παρά ε, βάση των 25.000 ε, ευρώ το μήνα. έτσι λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Υπήρχε βεβαιότητα το 2019 γιατί καθυστέρησε τον Brexit δύο φορές. Δεν είχαμε λοιπόν το ίδιο επίπεδο προσλήψεων μετά τις εκλογές το 2019 όπως έγινε στην περίπτωση άλλων βουλευτών. Ευχαριστώ. Uh, ε, δίνω τώρα το λόγο ε, στον κύριο Χαμεντού από την ΓΑΜΑ Επικοινωνίας. Για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω τι πρωτεύουσε του Κοινοβουλίου για το 2021 και τα δημοσιονομικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτές τις ε, προτεραιότητες, ε, καθώς όλα αποτελούν τους καρπούς των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Προεδρείο. Δεν θα μιλήσω για το ρόλο της ΓΑΜΑΔΑΛΤΑΚΟΜ, όλοι το ξέρουν. Εδώ είμαστε για να προσφέρουμε εξαντλητικέ πληροφορίε στου πολίτε, είτε απευθεία είτε μέσω των ΜΜΕ και προετοιμάζουμε και το έδαφος για τις δραστηριότητες επικοινωνίας των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών. Ε, όπως ε, ο Αντιπρόεδρος Σίλβα Περέιρα και οι Κούσα είπαν χτες, η επικοινωνία είναι μία από τις ε, θα είναι μία από τι κύριε προτεραιότητε ε, του Κοινοβουλίου για το 2021 και ελπίζω και για όλη τη θητεία. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι δυνατότητα να μπορούμε να ενημερώνουμε του πολιτε για το τι κάνει το Κοινοβούλιο, το έργο του και τον αντίκτυπο των αποφασεών του στην ε, ζωή των πολιτών ε, ή η πρόσθετη αξία που επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώ όλε οι δημοσκοπήσει μα λένε τώρα ότι έχουν μεγάλε προσδοκίε οι πολίτε από το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην προηγούμενη θητεία ε, είχαμε μεγάλη αύξηση της ικανότητάς μας ε, να απευθυνθούμε στους πολίτες μέσα από μεγάλο αριθμό πλατφορμών ε, ή μέσων, offline, online, ΜΜΕ, επισκέψεις, εκστρατείες, συμπράξεις, δραστηριότητες στα κράτη-μέλη. Δεν θα σας δώσω τώρα όλους τους αριθμούς όμως το Παρλαμεντάριο με ήδη το επισκέφτηκαν 7,5 εκατομμύρια άτομα, συγγνώμη 2,5 εκατομμύρια άτομα διορθώνω μιλητής. Στο Στρασβούργο ε, είχαμε μισό εκατομμύριο και 600.000 στο Βερολίνο, 130.000 στον ΣΥΝ και την πρώτη χρονιά, ένα εκατομμύριο επισκέπτες στις Βρυξέλλες το 2019, 300.000 στο Στρασβούργο, και σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ αυξήθηκε η παρουσία του Κοινοβουλίου εκθετικά θα συγκρίνει το 18 με το 19 θα ήταν λάθος λόγω των εκλογών όμως μπορώ να συγκρίνει το 2014 που είχαμε τις προηγούμενες εκλογές με το 19 ε, επί ήταν παρόν το Κοινοβούλιο στα ΜΜΕ το ε, 2019 σχέση με το 2014 5 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν τα ευρωπαϊκά ε, κτίρια το 2019. Είχαμε 3,4 εκατομμύρια φαν στο Facebook, 2 εκατομμύρια ακολούθηση στο Twitter. Όμως η πραγματική δοκιμή ήταν οι ευρωπαϊκές εκλογές. Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα αναφερθώ στη συνέχεια. Πιστεύω ότι καταφέραμε να έχουμε μια διαφορετική εκστρατεία που αναπτύχθηκε εσωτερικά από τις υπηρεσίες ε, καλούσε στην κινητοποίηση και στη συμμετοχή και ε, μας υποχρέωσε να γίνει μεγάλη προσπάθεια και επιγραμμικά αλλά μέσω και της κινητοποίηση των πολιτών στο ground game είχαμε ιδιαίτερα αποκεντρωμένη εκστρατεία, είχαμε συγκεκριμένους στόχους ε, κυρίως τους soft abstainers και τους νέους. Ε, φυσικά ε, τα αποτελέσματα ε, είναι 8,1% παραπάνω συμμετοχή. Μπορεί να μην σχετίζεται αυτό άμεσα με την εκστρατεία, αλλά μπορώ να σας αποδείξω στη συνέχεια ότι ήμασταν ένας από τους διάβλους, από τους φορείς που επέτρεψαν αυτή την αύξηση της συμμετοχής κυρίως ό,τι αφορά τους νέους. Ε, και για τα διδάγματα. Ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Ε, θα πρέπει να είναι μόνιμη. Δεν μπορούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες για το έργο του Κοινοβουλίου 6, 9, 12 μήνες πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας και ακριβώς ε, γι' αυτό στην προτεραιότητά μας για του χρόνου για το 2021 υπάρχει σημαντική αύξηση των πιστώσεων για τις εκστρατείες. Και ήδη έχει ξεκινήσει το 2020 με την εκστρατεία το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα και σε σχέση με την εκστρατεία για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, τη συζητήσαμε χτες, είναι το Europe Experience. Επίσης, ε, μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις που θα υπάρχουν αλλά νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία για το πόσο σημαντικό είναι να μένουμε κοντά στους πολίτες, κυρίως σε πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Και τα νούμερα που έχουμε και που αναφέραμε δείχνουν ότι πρόκειται για μια επένδυση που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επίσης, έχουμε σημαντικές επενδύσεις στα οπτικοακουστικά και έχουμε και επενδύσεις στους νέους, κυρίως μέσω της ε, οργάνωσης του European Youth Event. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και φυσικά όταν χρειάζεται μπορώ να έρχομαι για να συζητάμε πιο συγκεκριμένα από των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας παρακολούθησα με προσοχή. Πιστεύω ότι συνθετικά κάνατε μια σύνοψη. Παρουσιάσατε τις προτεραιότητες για το 2021, μιλήσατε για την εκστρατεία πληροφόρησης για τις επόμενες ευρωεκλογές που πρέπει να επεκταθεί σε βάθος χρόνου. Τα ποσά είναι τα αντίστοιχα. Ποιου είδους εκστρατεία τρία ή τέσσερα χρόνια πριν από τις εκλογές θα κάνουμε το 2021, δηλαδή η ουσία ποια θα είναι, το νόημα της εκστρατείας. Τώρα για τα κινητά στοιχεία του Παρλαμεντάριου. Να καταλάβω το μηχανισμό. Από πού θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα είναι άνθρωποι που θα έχουμε προσλάβει επιτόπου. Θα είναι ε, από τα σημεία επαφής που έχουμε. Θα ξεκινούν από τις Βρυξέλλες ή από το Στρασβούργο. Εκεί θα εκπαιδεύσουμε διαφόρους υπαλλήλους που θα εχουμε προσλαβει επιτοπου θα ειναι απο τα σημεια επαφης που εχουμε θα ξεκινουν απο τις βρυξελλες η απο το στρασβουργο εκει θα εκπαιδευσουμε διαφορους υπαλληλους που θα ταξιδεψουν σε όλη την Ευρώπη με το κινητό Παρλαμεντάριου. Είναι ένα αίτημα που υπέβαλα χθε και στο Γενικό Γραμματέα. Μιλήσατε για την επιτυχία του ε, European Youth Event, της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τους Νέους. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, λοιπόν, το ζήτησα χθε από το Γενικό Γραμματέα και σας το ξαναλέω. Να μας δώσετε μια αξιολόγηση του κόστους και να αναλάβετε τα έξοδα ταξιδιού, μετάβαση και στέγαση των νέων που έρχονται να συμμετάσχουν στο European Youth Event. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντούκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Σαστέλη, για την εκστρατεία την επικοινωνιακή για το 2021, να σας πω ότι σκοπός είναι να είμαστε σε φάση εκστρατείας για τα θέματα με τα οποία ασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας δεν θα επινοήσει θέματα, θα παρακολουθήσει αυτά που απασχολούν το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό το μήνα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η επικοινωνία στην εκστρατεία αντίστοιχα θα κινηθεί εκεί δεν θα εφεύρουμε δικά μας θέματα. Το 2021 θα κάνουμε σημαντική προσπάθεια για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και αν τελικά η διάσκεψη αυτή φέρει καρπούς και είναι επιτυχημένη και ε, ε, φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούν οι βουλευτές, τότε στα τέλη του 2022 θα είμαστε προς τα τέλη της νέας θητείας και θα κινόμαστε προς τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε καταβάλει σημαντική προσπάθεια online, θα έχουμε ενισχύσει τα ε, γραφεία σύνδεση στα κράτη-μέλη θα είμαστε όλο και πιο παρόντες στα μίντια, τα εθνικά και τοπικά μίντια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε γιατί πολύ συχνά τα περιφερειακά ΜΜΕ είναι πιο θετικά εναντί της Ευρώπης. Τώρα για, για τα μίνι παρλαμεντάριουμ, τα κινητά ε, το Europa Experience. Ποιοι υπάλληλοι θα μετακινούνται. Τρία είναι τα μοντέλα που θα ακολουθήσουμε. Κάποια στιγμή, σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι οι τοπικοί υπάλληλοι μας που θα το αναλάβουν αυτό, οι επιτόπου σε άλλες περιπτώσεις θα έχουμε τοπικούς ανθρώπους που θα έχουμε στρατολογήσει επί τόπου, γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό αυτό από το να στέλνουμε μονίμους υπαλλήλους να κάνουν το γύρο της Ευρώπης. Και έχουμε και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα σε, σε μια άλλη τρίτη κατηγορία περιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει το προσωπικό. Δηλαδή, ε, αν κάποιος μπαίνει να βιώσει ένα Europa Experience στη Λιουμπλιάνα ή στη, ε, στο Βερολίνο ή στην Κοπενχάγη θα καθοδηγείται από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι τρεις είναι οι άγουσες. Θα χρηματοδοτήσουμε ομάδες επισκεπτών, είτε το σύνολο των ε, εξόδων τους, είτε μέρος των εξόδων τους. Έχουμε γραμμή στο προπολογισμό για να βοηθήσουμε τις μειονεκτούσες ομάδες με κοινωνικά δίκτυα για οικονομικούς λόγους 54 ομάδες νέων θα χρηματοδοτήσουμε την επόμενη χρονιά με αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούμε ομάδες νέων που συμμετέχουν με δραστήριο και ενεργό τρόπο, δηλαδή που έρχονται και μας προτείνουν δραστηριότητες. Το 2020 άλλες 50 ομάδες θα χρηματοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο και έχουμε και τη χρηματοδότηση με το σπόνσορι, με τις χορηγίες, όπως χρηματοδοτούμε τις ομάδες επισκεπτών. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές μπορούν να επιλέξουν να στείλουν ομάδες επισκεπτών όχι μόνο στο, στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο για να δουν τις δραστηριότητες, αλλά για να συμμετάσχουν και ε, σε αυτό, με παρεμφερείς κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίντσιχ. Ναι, η εγκύτητα στον πολίτη είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, άρα λοιπόν αυτό το κινητό ε, παλαμετάριο με τα περισσότερα κινητά παλαμετάρια που θα υπάρχουν, πώς ακριβώς ε, θα κινούνται, δηλαδή θα μετακινούνται από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα, πόσο συχνά θα βρίσκονται σε κάθε κράτος και, και θα υπάρχει σχέση με αυτές τις υφιστάμενες εκθέσεις Europe Experience, δηλαδή τι θα ισχύει για τους ενδιαφερόμενους πολίτες οι οποίοι θα θέλουν να επισκεφθούν αυτές τις εκθέσεις, έτσι ώστε να Ρώσο και εγώ τους δικούς μας πολίτες. Ε, και ε, οι σχετικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα μέσα στα, στα κτίρια ε, της Ένωσης ή όχι. Τρία είναι τα διαφορετικά συστήματα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Στο Europa Experience το Προεδρείο αποφάσισε ότι πρέπει να υπάρχει ένα Europa Experience σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μέχρι το τέλος της θητείας. Είναι πραγματική προτεραιότητα το Europa Experience και αρκετά φιλόδοξο εγχείρημα. Είναι σαφές ότι δεν μένουν όλοι βεβαίως στις πρωτεύουσε τη χώρα μέλη, ούτε μπορούν όλοι να πάνε στην πρωτεύουσα τη χώρα τους. Και γι' αυτό θεσπίσαμε δύο άλλα συστήματα, role playing game mobile, δηλαδή μπορεί κανείς να παίξει το ρόλο ενός βουλευτή και άρα να το καταλάβει στην πράξη διαδικτυακά εδώ στο Παρλαμετάριο, για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, να καταλάβει πώ ακριβώ δουλεύουν οι βουλευτέ. και αυτό μπορεί να γίνει με κινητό τρόπο, δηλαδή σε συνεργασία με τα σχολεία, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τι ενώσει, του συλλόγου, τα δημαρχία, με διαφόρου φορεί δηλαδή που θέλουν να συνεργάζονται μαζί μα μέσω του γραφείου σύνδεση. και τρίτο στοιχείο, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα, και θα μπούμε στην πιλωτική φάση ε, εφαρμογής είναι το κινητό παρλαμεντάριουμ, είναι ειδική, ειδικό έτοιμο ε, δικό αίτημα του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουμε φορτηγά ή βανάκια που υπάρχουν και σε άλλες πολιτικές και μη πολιτικές δραστηριότητες φορτηγά, λεωφορεία, βανάκια που θα πηγαίνουν στην Ήπεθρο, στα χωριά στις περιοχές όπου δυσκολευόμαστε να οργανώσουμε δραστηριότητες δεν θα σταματήσουμε σε μια πόλη και θα ανοίξουμε την πόρτα του λεωφορείου έτσι απλά. Αντίθετα θα συντονιζόμαστε με δραστηριότητες που, ε, με τους τοπικούς φορείς και με τα τοπικά μας γραφεία σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή με τις συλλογικότητες του συλλόγους που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Και στο βαθμό του δυνατού θα έχουμε άμεση συμμετοχή βουλευτών. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Λίνα Λίνους από την Γενική Διεύθυνση Ίνλου, Υποδομών και Ελικοτανικής υποστήριξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που ε, μου δίνετε να ε, παρουσιάσω την δική μα ε, Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Ελικοτεχνική Υποστήριξη. Συνέχεια, βέβαια, τη παρουσίαση που έκανε ο Διευθυντή Σίλβα Περέρα και ο Γενικό Γραμματέα, αλλά και οι δύο αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα το πρωί. Πολύ σύντομα, να αναφερθώ σε αυτό που είπε και χθε ο Γενικό Γραμματέα, ότι δηλαδή στο πλαίσιο τη τελευταία βουλευτική θητεία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των όρων εργασία ε, τόσο των ευρωβουλευτών όσο ε, και του προσωπικού και στι τρει έδρε εργασία μα. Ε, και εφαρμόστηκαν αυτοί οι όροι εργασία με έμφαση σε όλε τι δραστηριότητε από την πλευρά τη Γενική Διευθυνσή ΕΝΛΟ. Συνεχίζουμε λοιπόν την ε, εφαρμογή αυτών των αξιών πολιτικής και στο πλαίσιο των νέων προτάσεων προπολογισμού που κάνουμε για το 2021. Ε, στη στρατηγική μας για τα κτίρια, σε σχέση με την οποία ο κύριος ε, Οσάκοφς έθεσε κάποια ερωτήματα, και ε, πράγματι το 2018 αποφασίστηκε λόγω στρατηγική και μπορούμε να σας την διαθέσουμε σε όλους μας και θα το κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες βασικές γραμμές, κάποιες βασικοί άξονες που διέπουν αυτή τη στρατηγική. Καταρχήν υπάρχει ε, μια γενική φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση. Δηλαδή σε όλες τις δράσεις προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και πάντοτε βασιζόμενοι στις υποδομές, ε, τις κτηριακές υποδομές και ε, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά ε, και στο πλαίσιο όλων των υπολείπων τεχνολογιών, για παράδειγμα παροχή υπηρεσιών ε, αυτοκινήτων ή για παράδειγμα χρήση πλαστικών μπουκαλιών στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου. Σε όλες λοιπόν μας τις πολιτικές εφαρμόζουμε αυτούς τους άξονες. Επίσης και στο πλαίσιο των επισκεπτών, στο πλαίσιο του Europa Experience, όπως ανέφερε μόλις τώρα ο συνάδελφος Ντουκυλιό, ότι προσπαθούμε δηλαδή και εκεί να εφαρμόσουμε τα της στρατηγικής και σε ό,τι αφορά και τις θέσεις στα τέσσερα στα οποία δεν υπάρχει ακόμα. Και συνεργαζόμαστε επίσης και με τη Γενική Διεύθυνση ε, Ασφάλειας, προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια των κτηρίων μας και προσπαθούμε να έχουμε διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών μας κτηρίων, έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το ε, χάσμα. Ε, που υπάρχει, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την απομόνωση δηλαδή του κτηρίου Τρεβδίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προπολογισμό, πολύ σύντομα το 2021, να σα πω καταρχήν προκατακτικά ότι ε, ποτέ δεν είναι γραμμικό ο προπολογισμό ε, τη γενική μα διεύθυνση. Δηλαδή, παρέχουμε υπηρεσίε σε άλλε υπηρεσίε και χρησιμοποιούμε πολλέ δημοσίε συμβάσει ουσιαστικά αποκλειστικά δηλαδή έχουμε 600 συμβάσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ε, ε, υπάρχουν αλλαγές, δυναμικές αλλαγές στην αγορά και υπάρχει αυξομοίωση των τιμών. Και αυτό λοιπόν το λέω για να απαντήσω στο ερώτημα που ήδη έθεσε ο κύριος ε, Μπόζεν Λάγκερ. Δηλαδή ότι αυξομοιώσεις εδώ στις ενεργειακές τιμές πηχούν ακριβώς τις μεταβολές στις τιμές εδώ στις Βρυξέλλες. Είχαμε δηλαδή αύξηση κατά 28% ενώ στο Λουξεμβούργο για παράδειγμα μπορέσαμε να μειώσουμε ε, το, τη σχετική δαπάνη ε, λόγω του, ε, της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας, αυτοδύναμης δηλαδή γεωθερμικής ενέργειας ε, στο κτίριο Αντενάουαρ. Άρα λοιπόν πρόκειται εδώ για ένα προπολογισμό ο οποίος προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς. Επίσης ε, πρόσφατα υπήρξε μια μείωση στο ε, προπολογισμό μας, όπως ανέφερε ο κύριος ε, Κλέτη, με αποτέλεσμα 236 εκατομμύρια ευρώ σε χρήση κατά 99% εκτέλεση δηλαδή του προπολογισμού μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι στιγμής αξιοποιούμε σχεδόν στο άκυρο απόλυτα τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και βέβαια ακολουθούμε τα όσα προβλέπει η ε, ε, ε, ενεργειακή οδηγία, δηλαδή ε, τις ε, των κτηρίων ετησίως. Επίσης έχουμε τα όσα, έχουμε, τα όσα έχουν προσθεθεί βασίζονται και στα, στα νέα κέντρα Europe Experience αλλά και στις ανακοινήσεις οι οποίες έχουν εμ, εγκριθεί ε, με βάση βέβαια και την Γενική Διευθύνση Προπολογισμού δηλαδή και το κτίριο ΣΠΑΚ αλλά και την κατασκευή όπως είπαμε του εκτήριου Adenauer στο Λουξεμβούργο. Αυτά λοιπόν είναι τα ε, κύρια στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε κάποια αύξηση του προπολογισμού 14,2 δηλαδή εκατομμύρια αύξηση σε σχέση με το 2020 δηλαδή 6,3% αύξηση της ε, πρότασης προπολογισμού μας. Δηλαδή 240,72 ε, εκατομμύρια ευρώ η πρόταση προπολογισμού. Κύριε Σαστέλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για τους χώρους Europa Experience, όπως έκανε και ο συνάδελφος από την DG.com. Για εσάς είναι πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση το κτηριακό γιατί υπάρχει και αυτή η προθεσμία να μεταφέρουμε σε όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος του 2021 αυτή την, αυτό το εγχείρημα για το Europa Experience. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τη λογική με τις συμβάσεις των τοπικών γραφείων. Πόσα τοπικά γραφεία θα μετασχηματιστούν, θα μετεγκατασταθούν, θα τελείξει η σύμβαση. Ποια λογική έχετε ακολουθήσει σε κάθε πρωτεύουσα γενικά. Ευχαριστώ κύριε Λίνος. Ευχαριστώ Α, πολύ. Πρόεδρε, αυτή είναι μια πολύ εύστοχη ερώτηση, η οποία είναι εύκολη αφενό στο να απαντηθεί, αλλά και δύσκολη. Καταρχήν να πω ότι συνεργαζόμαστε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ουσιαστικά συνεργαζόμαστε ω εταίρεια, έτσι ακριβώ λοιπόν να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση του ε, Προεδρού και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πραγματικότητα υπάρχουν γραφεία επικοινωνία και επαφή, ε, δηλαδή σύνδεσμοι σε 36 ακτέ, σε πρωτεύουσε ε, ενό. Σε ορισμένα από τα κράτη-μέλη υπάρχει και ένα δεύτερο γραφείο επικοινωνία. Τώρα, ε, το Προεδρείο ζητάει να έχουμε σε, όλα αυτά τα γραφεία του Europa Experience, που καταρχήν προφανώς εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στασβούρο και από εκεί και μετά στο Βερολίνο, στο και ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο εκεί, στη Λουμπλιάνα, στην Κοπενχάγη και στο Ταλίν που θα ανέξει τώρα, ε, στο εγγύς μέλλον. Και σε ό,τι αφορά ε, ορισμένε άλλε πρωτεύουσε, έχουμε δει ότι η μίσθωση ορισμένων ακτηριακών εγκαταστάσεων γραφείων, δηλαδή εκεί που έχουμε, ε, έρχεται προς, κοντεύει στο τέλο, σε ό,τι αφορά τα σχετικά δηλαδή στο τρία συμβόλαιο, και γι' αυτό ε, προβλέπουμε να έχουμε δημόσιου χώρου ε, για το ε, Europe Experience, αλλά και για την εγκατάσταση των γραφείων του προσωπικού του Κοινοβουλίου, αλλά και του προσωπικού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί. Αυτό λοιπόν, αυτά τα συμβόλαια φτάνουν προς το τέλος μας δίνουν κάποια ευελιξία και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο δηλαδή να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητε που έχουμε σε διαφορετικές πρωτεύουσε. Και βέβαια ε, πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι η δυναμική εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, ε, τιμές ε, μίσθωσης ε, των, αυτών των εργαστάσεων είναι τελείως διαφορετική από ό,τι πριν από 25 χρόνια και το λαμβάνουμε λοιπόν και αυτό υπόψη μας. Αυτά σημαίνουν στο Δουβλίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Πράγα στη Στοχόλμη και στη, στη Χάγη, ενώ πολύ σύντομα θα υπάρξουν και εννέα ακόμα σημαία μέσα στο 2021 πια όπου θα συμβούν ε, πολλά δηλαδή ταυτόχρονα. Ε, και εκτιμώ τα σχόλια που έγιναν ε, χθες από την πλευρά διαφόρων ευρωβουλευτών, μεταξύ αυτών και από την πλευρά τη κυρία Κέλλερ, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα και για τα ε, κράτη-μέλη της και Ανατολικής Ευρώπης να ανοίξουν περισσότερα τέτοια κέντρα έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες για να περάσουμε ακριβώς τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτά τα τέταρτο Europe, Experience. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν άλλα σχόλια, ερωτήματα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αλήνους για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια ερωτήματα που έθεσα χθε στο Γενικό Γραμματέα. Ήταν τεχνικά ερωτήματα και ο Γενικός Γραμματέας δεν μπόρεσε να απαντήσει. Κυρία Γενική Διευθύντρια, σας ρώτησα για το θέμα της συντήρησης των κτηρίων και είχαμε καταλάβει τη σημασία τους γιατί επισκεφθήκαμε αυτά τα κτίρια. Υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή, δεν τη βρίσκω στο, στο τμήμα 2. Είμαι νεοφώτιστη βέβαια και μαθαίνω σιγά σιγά να διαβάζω τους πίνακες. Στον πίνακα για τις επενδύσεις, για τις σημαντικές επενδύσεις, για τη μόνος, η της στέγης, για θέματα θεμελίων, πράγματα που δεν, δεν είναι πολύ ωραία τα άλλα, είναι σημαντικά γιατί. Ε, για την ε, ε, σωστή ύπαρξη των ε, κτηρίων, τη σταθερότητά τους. Και έχουμε και το 3% των δαπανών. Για το κτίριο Σπινέλη, είχαμε επισκεφθεί και είδαμε σημαντικές εργασίες στους ηλεκτρολογικούς μετασχηματιστές, τους καυστήρες και το καθεξής. Και είχα θέσει και το ερώτημα για το Poland Risk 10,2 εκατομμύρια ευρώ είναι εγγεγραμμένα στο προϋπολογισμό στο τμήμα 2. Μήπως μπορείτε να μας τα εξηγήσετε καλύτερα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγγέλα για αυτά τα ευστοχά ερωτήματα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά ε, το κόστος συντήρησης ε, και την ανακαίνιση ε, κτηρίων, είτε δηλαδή των ίδιων των κτηρίων, είτε τα τεχνικά ε, δηλαδή, για παράδειγμα ε, διαχείριση του συνολικού του κριτήριου, για παράδειγμα διαχείριση του συστήματος Ε, καταρχήν έχουμε ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, ανακαίνιση ε, το οποίο καλύπτει όλα τα κτίρια, δηλαδή και αυτά του Στρασβούργου και αυτά των Βρυξελών. Και έχουμε εδώ και ένα δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα. Και αυτά τα, αυτές οι δαπάνες δηλαδή ανακαίνησης και επενδύσεων περιλαμβάνονται στη γραμμή 2007. Και βέβαια, θέλετε, μπορούμε να ε, δούμε διμερώς αυτές τις ε, ε, γραμμές για να μην σπαταλήσω όλο το χρόνο εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η γραμμή αναφέρεται ακριβώς στην, στην, εγκατάσταση εκ των υστέρων περαιτέρων συστημάτων. Ενώ στην 2022 έχουμε να κάνουμε με γενικότερα ζητήματα συντήρησης και καθαριότητας ε, και ε, στις τρεις έδρες εργασία ε, του Κοινοβουλίου στα όλα τα σχετικά κτίρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κτίριο ΣΠΑΚ, ελήφθη μια απόφαση από το Προεδρείο τον Ιούλιο του 2018 να λάβει χώρα ένας διαγωνισμός αρχιτεκτονικός έτσι ώστε να υπάρξει μια ανακαίνιση εκβαθέων προκειμένου να καταστεί πιο ε, φιλοπεριβαλλοντικό αυτό το κτίριο ή ε, εναλλακτικά για να ανακατασκευαστεί ε, το κτίριο. Και όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο αρχιτεκτονικός αδιαγωνισμός, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Προεδρείο και το Προεδρείο με τη σειρά του θα αποφασίσει ε, ποια από αυτές τις δύο εναλλακτικέ θα επιλέξει. Δηλαδή αν θα υπάρξει αυτή η ανακαίνιση, η ριζική ανακαίνιση προκειμένου να γίνει πιο φιλοπεριβαλλοντικό το κτίριο ή η ανακατασκευή του. Και βέβαια εσείς ε, θα ε, παραμένετε ενήμεροι από τη δική μας πλευρά. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως γιατί ζητούμε εδώ να λάβουμε προπαρασκευαστική χρηματοδότηση. Γιατί και οι δύο αυτές εναλλακτικέ είναι πολύ σημαντικές. Οπότε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι τεχνικές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα ε, το κέντρο δερμηνέας, για παράδειγμα, για την οργάνωση της Γερμανίας ε, που βρίσκεται σε μια μεγάλη αίθουσα στο κτίριο ΣΠΑΚ να έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο κτίριο. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, τις θέσεις συνεδριάσεων των ε, δημοσιογράφων, τα press centers ε, αλλά και τις θέσεις συνεδριάσεων σε ό,τι αφορά το Προεδρείο αλλά και τη διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή τις σχετικέ αίθουσε συνεδριάσεων για αυτά τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, όλα λοιπόν, όλες αυτές οι αίθουσες θα πρέπει φυσικά να εγκατασταθούν αλλού ε, ε, όποια και αν από τι δύο εναλλακτικέ επιλεγεί για το κτίριο ε, ΣΠΑΚ. Οπότε από τώρα θα πρέπει να προβλέψουμε αυτέ τι δαπάνε. Και από εκεί και μετά, βέβαια, ο σχεδιασμός, ο αρχικός σχεδιασμός για το ΣΠΑΚ ήδη χρήζει κάποιων πρώτων κονδυλίων και γι' αυτό έχουμε ζητήσει αυτά τα 2,3 συμπληρωματικά εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο ε, Βάλτερ και από την ε, Γενική Διευθυνσή Τράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για την γάμα δελτα μετάφρασης. Θα ξεκινήσω με κάποιους στόχους ε, στρατηγικούς για τη δική μας δουλειά. Και όπω λέει και το ίδιο το όνομα, είναι να είμαστε ε, ουσιαστικά εντός της πολυγλωσσίας να χρησιμοποιούμε και τις 24 γλώσσες στην Ήπειρό μας ε, και να παράγουμε μεταφράσεις ε, νομοθετικού και μη νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά ο δεύτερος στόχος που θέλω να τονίσω είναι να επικεντρωθούμε στην καθαρή γλώσσα. Αυτό είναι ο νέος στρατηγικός στόχος ή τη γλώσσα των πολιτών όπως την αποκαλούμε. Και ταυτόχρονα να είμαστε και αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Έχοντας αυτά κατά νου, Επίσης ε, είδαμε ε, ποια είναι τα περιουσιακά μας στοιχεία στην γάμα μετάφρασης. Καταρχήν ε, είναι η γλωσσική αρχή στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά συνεργαζόμαστε εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα αλλά και με φορείς σε εθνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία που έχουμε και που αναπτύσσουμε και στην οποία επενδύουμε τα χρήματα. Επίσης, τεχνητή νοημοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούμε να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε και για τις 24 ε, γλώσσες. Δηλαδή, οι γλώσσες ε, που μιλώνται λιγότερο θέλουμε να τις βάλουμε σε ένα ψηφιακό χάρτη. Αυτό είναι το καθήκον μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι ε, άνθρωποι. Μιλάμε για πάνω από 1.100 ε, εμπειρογνώμονες ε, στην διευθυνσή μας, ε, ομαδοποιούνται σε τρεις διευθύνσεις. Αυτοί που ασχολούνται με τη μετάφραση, αυτοί που ασχολούνται με την υποστήριξη στη μεταφραστική διαδικασία και αυτοί που ασχολούνται με τους πόρους. Μπορεί να ακουστεί πολύ εντυπωσιακό το output όταν ε, πω 2,5 εκατομμύρια σελίδες ε, το χρόνο, όμως αυτό ισχύει για το 2018 που είχαμε πολλές εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά μέσο όρο μιλάμε για 2 εκατομμύρια σελίδες ή παραπάνω. Αν δούμε τα νούμερα του 2018, μπορώ να τα συγκρίνω με τα 7 βιβλία του Χάρι Πότερ. Αν ε, πάρουμε και τα 7 βιβλία του Χάρι Πότερ και τα μεταφράζουμε σε 23 γλώσσες ε, κάθε δύο εβδομάδες ε, για ολόκληρο το χρόνο. Αυτός είναι ο αριθμός των σελίδων που μεταφράζουμε στη διευθυνσή μας. Από τη σκοπιά αυτή, μιλήσαμε για την πρόταση του προπολογισμού 2021 θέλουμε καταρχήν να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογία και θέλουμε να αναπτύξουμε τεχνολογία που να υποστηρίζει μια συνεκτική μετάφραση της νομοθεσίας καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας και δεύτερον να αναπτύξουμε τεχνολογία που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε αυτό που λέμε μια καθαρή γλώσσα, απλή γλώσσα, τη γλώσσα των πολιτών. Δεύτερο, γραμμή του προπολογισμού αφορά την τεχνολογία που θα μας βοηθήσει στο θέμα της αποτελεσματικότητας. Κάτι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια καθήκοντα αυτόματα, αλλά και να έχουμε ένα χαρακτηριστικά όπως το μετάφραση του λόγου σε κείμενο ή την αναγνώριση φωνής. Παραδείγματο χάρη, καλύτερη προσβασιμότητα στις συζητήσεις για τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής. Αυτό μπορεί να εισαχθεί πάρα πολύ γρήγορα και για τους βουλευτές αλλά και για τους πολίτες. Η τρίτη επένδυση θα αφορά την κατάρτιση των ε, υπαλλήλων ε, στα νέα αυτά καθήκοντα για να αναπτύξουν ε, ουσιαστικά να προωθήσουν τη χρήση αυτής της γλώσσας των πολιτών σε όλα τα στάδια και για όλους τους συντάκτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να κλείσει αυτό το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, παρόλο που είναι δύσκολη διαδικασία, ανυπομονούμε να τη θέσουμε σε εφαρμογή σας. Ευχαριστώ και τον προτέρων για την υποστήριξή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Σαστέλ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντα. Θα απευθυνθώ σε εσά ε, για να σας ευχαριστήσω ε, για το έργο των μεταφραστών και των ε, διαρμηνέων. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τη σύμπραξη καινοτομία που η δική σα Γενική Διεύθυνση θέλει να υλοποιήσει. Μα ε, λέτε ε, ότι οι κοινοβουλευτικέ ε, συζητήσει σε πολλέ γλώσσε θα μεταγράφονται αυτόματα. Θέλω να δω ποιο είναι το κόστο ολόκληρου αυτού του προγράμματος και ε, θέλετε ουσιαστικά προοδευτικά να το στην ε, δομή πληροφορικής του Κοινοβουλίου και για ποια χρήση. Είναι κάτι σημαντικό. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το κόστος ενός μέρους των μεταφράσεων που έχουν να κάνουν με τις επεξηγήσεις ε, ψήφων. Ε, ρώτησα και χθε το Γενικό Γραμματέα για το θέμα αυτό πέρσι στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια συζήτηση είχαμε ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα να μας πει σε νούμερο ποιο είναι το κόστος των επεξηγήσεων ψήφου και μας είπε τότε ότι κοστίζει 29.400 ευρώ, δηλαδή πάνω από 900.000 ευρώ το χρόνο, 21.400 ευρώ την ημέρα και ουσιαστικά ε, θα ήθελα ε, να ξέρω αν είναι σκόπιμες αυτές τις επεξηγήσεις ψήφου μου. Επιβεβαιώνετε εσείς αυτό το νούμερο και θα θέλαμε να μου πείτε τι κοστίζουν οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για την σύμπραξη καινοτομία. Είναι όντω ε, κάτι καινούριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλα θεσμικά όργανα ακολουθώντας δυνατότητες που έχουμε στο δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα το speech to text είναι κάτι που, όπως σας είπα και πριν, μπορεί να συνδεθεί με νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να προσφερθούν κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ή σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των μελών του Κοινοβουλίου, γιατί θα μας επέτρεπε να έχουμε αυτόματη μεταγραφή των ζωντανών συζητήσεων. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Μπορεί να συνδεθεί και θα συνδεθεί και με την ε, μηχανική μετάφραση, machine translation, που θα μπορούσε να ε, ενταχθεί στο σύστημα, αλλά αρχικά θα ξεκινήσουμε μόνο με τις ολομέλειες και μόνο για λίγες γλώσσες ε, και στη συνέχεια θα το διευρύνουμε αυτό και σε υπόλοιπες συνεδριάσεις και γλώσσες. Ο βασικός στόχος είναι για την προσβασιμότητα ε, των κοφών και των ατόμων με προβλήματα κοής. Ο στόχος είναι να δώσουμε την ευκαιρία όλες οι γλώσσες να αναπτυχθούν σε αυτό το σύστημα γιατί η εμπορική αγορά δεν είναι απαραίτητο ότι θα παράσχει τα ίδια στοιχεία και για τις 24 γλώσσες, καθώς κάποιες ε, μιλούνται λιγότερο και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι καθήκον μας αυτό κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε κάποιες ε, γλώσσες στο ψηφιακό χάρτη, αλλά και να δώσουμε περαιτέρω εγγύησεις ε, της πολυγλωσσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και εκτός. Ε, το εκτιμόμενο κονδύλιο, το εκτιμόμενο κόστος είναι ένα εκατομμύριο ένα έτος για μία τριετή περίοδο της καινοτόμου σύμπραξης με τον επιλεγμένο εταίρο. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το κόστος και αυτό δεν έχει ακόμη υπολογιστεί τη ε, ε, επένδυσης επιτόπου, δηλαδή όσων θα συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη. Είναι λοιπόν πολύ σκόπιμη η ερώτησή σας γιατί πρώτη φορά θα το κάνουμε αυτό και γι' αυτό η Διευθύνουσα Επιτροπή θα συμπεριλάβει όλες τις γενικές διευθύνσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου που ενδιαφέρονται για αυτές τις υπηρεσίε Για να σας πω ένα παράδειγμα, πριν του χάρη την Προεδρία, την Ολομέλεια, τους διερμηνείς, πολλού άλλους που θα χρησιμοποιήσουν αυτέ τι υπηρεσίε. Επίση, επομένω, η γάμα δέλτα είναι ο κεντρικό κόμβο για αυτό το σχέδιο για αυτό το πρόγραμμα καινοτόμου σύμπραξη. Είναι το πρώτο έτος που εφαρμόζεται, αλλά αυτή η αρχιτεκτονική αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό. Για την δεύτερη ερώτησή σας, για την Ολομέλεια, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επεξηγήσεις ψήφου και τις προφορικές τροπολογίες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε το πρώτο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, η μετάφραση γίνεται κατόπιν αιτήματο. Δεν υπάρχει αυτόματη μετάφραση. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει αίτημα, τότε μεταφράζεται. Αυτό είναι δύσκολο λοιπόν να το προβλέψουμε στον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Αν όχι, να δώσω το λόγο στην κυρία Νιέσκα Βαλτεντρόπ από την ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΛΙΝΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω την ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ ΛΙΝΚ που είναι υπεύθυνη για την επιμελητία και για τη διερμηνία τι κάνουμε, παρέχουμε γλωσσική, τεχνική και πολιτική υποστήριξη για τη διοργάνωση ε, συναντήσεων και διάσκεψεων ε, σε καθεστώς πολυγλωσσίας καθώς ε, και άλλων εκδηλώσεων όπως οι εκθέσεις των βουλευτών. Μέσω αυτού βοηθάμε να προωθήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων, καθώς διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των μελών ε, και την νομοθετική διαδικασία, αλλά και την απεύθυνση στους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είμαστε μαζί σας από τη στιγμή που θέλετε να οργανώσετε τη συνεδρίασή σας. Έχουμε διοργανωτές ε, των συναντήσεων και συντονιστές ε, των εκδηλώσεων όταν κλείνεται την συνεδρίαση οι κλητήρες μας ε, σας βοηθούν με το να υλοποιηθεί το έργο των Επιτροπών και των λοιπόν φορέων. Επίσης ε, είμαστε εκεί και παρέχουμε τις ε, τεχνικές διευκολύνσεις, παρέχουμε τους τεχνικούς και τις τεχνικές επιδομές και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, παρέχουμε την διερμηνία με διερμηνείς που εργάζονται in situ σε ταυτόχρονη μετάφραση, αλλά σε συνοδεύουν και στις αποστολές. Έχουμε προσωπικό 550 ατόμων και κατανέμονται σε τέσσερα τμήματα και με περηφάνεια λέμε ότι η διαχειριστική μας ομάδα, οι διευθυντές μας είναι κατά 70% γυναίκες σε συνολικό πληθυσμό 58% γυναικών που είναι παρούσες. Να αναφερθώ την ε, ε, βιώσιμη μετάφραση σε πλαίσιο πολυγλωσσίας ε, σε κάθε συνεδρίαση το 2018 που είναι το έτος αναφοράς είχαμε περίπου 7.000 συνεδριάσεις με διερμηνία με 250 μόνιμο προσωπικό και περίπου 1.500 freelance που εργάζονται στις ίδιες ομάδες και αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις ε, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στη διατηρήση της αγοράς, γιατί ε, ουσιαστικά πιστοποιούμε τους διερμηνείς μας μαζί με άλλα θεσμικά όργανα, μαζί με την Κομισιόν και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είμαστε σε ηγετική θέση σε αυτή την παροχή υπηρεσιών, ο διοργάνωση συνεδρίας. Ε, δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 24 γλώσσες που να μεταφράζονται. Επίσης, αυτό απαιτεί επενδύσεις, ε, ε, ίδιοι διερμηνείς πρέπει να αναπτύξουν ε, τα δεξιότητές τους, να διατηρήσουν τις γλώσσες τους, πρέπει να υποστηρίζουμε τα πανεπιστήμια και τη νέα γενιά των ατόμων που συνεργάζονται μαζί μας. Όμως χρειάζεται και πολύ σημαντικός προγραμματισμός και πρόσληψη μαζί με το ε, γραφείο μας, ε, με το προσωπικό που είναι στα γραφεία και την ανάπτυξη software. Και μπορώ να πω ότι μαζί με την Κομισιόν τώρα εξετάζουμε τι γίνεται με τα εργαλεία μας, την τεχνολογία των πληροφοριών, προκειμένου να βελτιώσουμε τα εργαλεία για την πρόσληψη. Το δεύτερο τμήμα των ε, δραστηριοτήτων μας ε, και αυτό καλύπτει τα πάντα, είναι οι υπηρεσίες ε, διοργάνωσης συνεδρίων. Το 2018, για να σας δώσω κάποια στοιχεία, είχαμε πάνω από 23.000 συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο. Βρισκόμαστε εκεί, όπως σας είπα, Είχαμε επίσης, επίσης μάλλον 250 με 300 εκθέσεις ε, διοργανώνουμε κάθε χρόνο και οργανώνουμε και τις συναντήσεις ε, της Ενδρίας των Πολιτικών Ομάδων ε, πέρα από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτά έχουν προβλεφθεί στον προπολογισμό για την διοργάνωση συνεδρίων. Επενδύουμε μαζικά στην καινοτομία αναπτύσσουμε την έννοια της οργάνωσης των Stop Conference. Ε, τώρα ε, έχουμε ε, το εργαλείο για να έχουμε μία συγκεκριμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση των εγγραφών και αυτό θα συνδεθεί και με το σύστημα επιστοποίησης της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ SAFE. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, υπηρεσίες remote και για webinars ε, και ε, για διάφορες συνεδριάσεις και τέλος πρέπει να εξυγχρονίζουμε συνεχώς την υποδομή μας και έχουμε γραμμή του προπολογισμού 10 εκατομμύρια για το σκοπό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαστέλ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ανια Βάλτερ Ντρόπ, να σας θέσω ένα ερώτημα για τα τελευταία σας λόγια, για τη στρατηγική εξυγχρονισμού των υποδομών για τις διασκέψεις και τις συνεδριάσεις μας. Μπορείτε να σταθείτε λίγο παραπάνω στο θέμα αυτό. Μιλούμε για τηλεδιάσκεψη τελευταίας γενιάς με κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη στρατηγική, για την ουσία αυτή της στρατηγικής αλλά και το κόστος που συνεπάγεται. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πράγματι, είναι μια στρατηγική που βασίζεται σε απόφαση του Προεδρείου. Επιδιώκουμε να πετύχουμε συνέργειες και να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί και υπάρχουν στο, στην αγορά. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στην έκθεση την εμπορική του Άμστερνταμ ε, και είδαμε τι μπορεί να μας χρησιμεύσει ως εργαλείο για να στηρίξουμε τις διασκέψεις, τις συνεδριάσεις, τις συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όντως, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε συνέργειες. Το μοναδικό σημείο συντονισμού Πώς θα συγκεράσουμε δηλαδή όλες τις τεχνολογίες στις αίθουσες συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεδιάσκεψης. Ξέρετε, όλα αυτά τα διαχειρίζονται διαφορετικά μέρη, διαφορετικά τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής εξαρτώμαστε πολύ και από το δικό τους προϋπολογισμό και από το κατά πόσο εκείνοι μπορούν να αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής με βάση τον προϋπολογισμό που έχουν. Και πέραν της τηλεδιάσκεψης που αναφέρατε, οι διερμηνεί μα, οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ στην αίθουσα, εξαρτώνται από τα δίκτυα πληροφορική και τα πληροφορικά εργαλεία που έχουμε, γιατί σε τέτοιου είδου συνεδριάσει πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία εξετάζονται από την εκάστοτε επιτροπή, από την επιτροπή σας εμπροκειμένου. Τώρα, το συνολικό κόστος κατανέμεται ε, σε διάφορες γραμμές. Υπάρχει μια γραμμή προϋπολογισμού για τα αποκεντρωμένα έργα ανάπτυξης και σχεδιασμού δράσεων πληροφορικής. Είναι μια νέα γραμμή στο προϋπολογισμό για την οικονομική χρήση 2021 Μιλούμε για 1.200.000 ευρώ για την ανάπτυξη νέων εργαλείων όπως αυτά που ανέφερα. Π.χ. τα εργαλεία για να υποστηρίξουμε τη δημιουργία webinar διαδικτυακών σεμιναρίων ή αντιστοίχων τέτοιων δράσεων και εφαρμογών. Έχουμε και άλλες πιστώσεις 214.000 ε, ευρώ για ε, τον εξοπλισμό των θουσών και τον ε, εξοπλισμό και την εκπαίδευση των τεχνικών. διότι οι αίθουσες ελέγχονται τεχνικά από ένα ε, κέντρο διοίκησης, τεχνικής διοίκησης, με κεντρικό τρόπο και όχι μόνο από τον τεχνικό που είναι παρόν στην αίθουσα. Και θέλουμε και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής ε, από μακριά. Δηλαδή υπάρχουν αίθουσες συνεδριάσεων οι οποίες είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, συμμετέχοντες οι οποίοι δεν βρίσκονται στην αίθουσα αλλά παρακολουθούν με ηλεκτρονικό οπτικό ακουστικό τρόπο και πρέπει να τις αυτές. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Είδα να δώσω το λόγο στον κύριο Βάλτερ Πετρούτσε από τη Γενική Διεύθυνση ITEC πληροφορικής. Ο κύριος Πετρούτσε είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Να σας παρουσιάσω εν συντομία τη γενική μας διεύθυνση, η οποία δίνει στήριξη σε θέματα πληροφορικής και δημοσίευσης ε, για τα μέλη του Κοινοβουλίου, τους βοηθούς και το προσωπικό, συντηρεί και ανα... τις ηλεκτρονικές υποδομές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ε, επικουρεί στο διοικητικό έργο και κάνει λειτουργίες εκτύπωσης ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή μετασχηματιζόμαστε μαζικά για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίε που προσφέρουμε παραμένουν καινοτόμε, ασφαλεί και προσαρμοσμένε και προσαρμοζόμενε στι εξελισσόμενε ανάγκε των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προσωπικού. Θέλουμε μια εσωτερική δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθεί κατά πόδα στις τεχνολογικές εκτελήξει. Θέλουμε να έχουμε τεχνολογία εχμής για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το προσωπικό και τη διοίκηση και για να γίνει αυτό τρεις είναι οι γραμμές δράσης που ε, ακολουθούμε. Στην πρώτη γραμμή δράσης Θέλουμε το οικοσύστημα πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι έτοιμο για το μέλλον και γι' αυτό χρειαζόμαστε 4,2 εκατομμύρια για το cloud και το data center, 2,6 εκατομμύρια για τα data hybrids και 3,5 εκατομμύρια για την κυβερνοασφάλεια. Το 2021 θα είναι κρίσιμη χρονιά για την επέκταση της αρχιτεκτονικής δομής στο cloud, νέες τεχνολογίες όλο και περισσότερο νέες ε, τεχνολογίες λειτουργούν μόνο στο cloud και όχι εκτός αυτού και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην αποκοπεί από ε, το ηλεκτρονικό νέφος, από το cloud. Αυτές οι τεχνολογίες θα αυξήσουν τη δυνατότητά μας, την αντοχή μας, την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών πληροφορικής. Και έτσι θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη, με γρηγορότερα, με ασφαλή τρόπο, με στέρεο τρόπο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τα data ε, centers μπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι τα data center είναι ε, ε, ευαίσθητα και πρέπει να παραμείνουν εντό των εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχει απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών μα data center και του cloud ε, πρέπει να έχουμε του απαραίτητους πόρους και γι' αυτό ζητούμε αυξημένο προϋπολογισμό για το 2021 και η αύξηση έχει ως σκοπό να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει στο έπακρο και του δύο κόσμου και το cloud και τα data center. Και πρέπει να έχουμε και επαρκή εσωτερική ικανότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια ε, των θεσμικών μας οργάνων. Οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται όλο και πιο προηγμένες και συνεχώς πρέπει να αναβαθμίζουμε την ικανότητά μας. Έχουμε έτοιμα για 3,5 εκατομμύρια ευρώ στο προϋπολογισμό, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των αναγκών μας, αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο μπορούμε να φέρουμε σε πέρας. Ε, αντιστοιχεί στη διοικητική ικανότητά μας να ε, να είμαστε επαρκή σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Έχουμε και τους υβριδικούς υπολογιστές και πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπους και σε, αυτό, σε αυτή τη τεχνική υποδομή με πιο, πλήρη και πιο, πιο πλήρης και πιο κινητές συσκευές για όλους, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε ανα πάσα στιγμή. Μιλούμε για ένα κινητό περιβάλλον εργασίας και αυτό τονίζεται από το ε, περιβάλλον χωρίς εκτύπωση, δηλαδή ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς πάρα πολλές εκτυπώσεις, χωρίς ε, μεγάλη εκτύπωση χαρτιού για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Είχε ήδη ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και θα επεκταθεί και τα επόμενα χρόνια. Και έτσι ε, θα καταπολεμήσουμε και την απαξίωση των σταθερών υπολογιστών γραφείου. Έχουμε αυξημένο, αυξημένα αιτήματα για νέες υπηρεσίες. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και για να δώσουμε λύσεις στα μέλη και στη διοίκηση οριστικές. Δεν θα αναπτύσσουμε δηλαδή εφαρμογές από μόνοι μας, γιατί αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο ε, και ε, ε, δεν είμαστε αποτελεσματικοί σε άμεσο χρόνο, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε άμεσα τα αιτήματα των μελών και γι' αυτό θα αγοράζουμε έτοιμα πακέτα από την αγορά. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε τις υφιστάμενες ε, υποδομές εκεί όπου υπάρχει απαξίωση των συσκευών. Μιλούμε για διοίκηση, για διαχείριση της απαξίωσης Πρέπει να αντικαταστήσουμε το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το οποίο γυράσκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις αίθουσε συνεδριάσεων. Υπάρχει ένα έτοιμο υποκατάστατο που θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2021 σε όλες τις αίθουσε όπου υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις Βρυξέλλες και το 2022-2023-2024 θα αντικαταστήσουμε το παλαιότερο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ε, για τις δύο έδρες, και για το Βρυξέλλες και για το Στρασβούργο. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριο Σαστέλ, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Είχα κάποιε ερωτήσει να σα θέσω. Η παρουσίασή σα όμω ήταν σαφή και ήδη απάντησε σε κάποιες από τις ερωτήσεις για την κυβερνοασφάλεια π.χ. και την τεχνολογική εξέλιξη. Βλέπω ότι για εσά είναι σημαντικό αυτό το διακύβευμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι και το κατανοούμε. Ειδικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο έχει επαξιωθεί και προγραμματίζεται να το αντικαταστήσετε. Επίσης αναπτύσσετε ε, υβριδικούς μηχανισμούς και συσκευές. Για τέτοιου είδους μηχανισμούς μπορείτε να μας ποσοτικοποιήσετε την κατάσταση, γιατί πρέπει να δούμε ε, και υπό αυτή την οπτική γωνία ποια εξοικονόμηση θα κάνουμε εάν τελικά υπάρχει βρεδικό μηχανισμός που θα αντικαταστήσει και το κινητό και το σταθερό υπολογιστή και όλα τα άλλα τεχνολογικά μέσα που ε, χρησιμοποιούμε σήμερα. Oui, monsieur le rapporteur, merci pour euh, cette question. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, κύριε εισηγητά. Πράγματι, θέλουμε να αναπτύξουμε υβριδικού υπολογιστές πανίσχυρους που θα μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε σε κίνηση με σκοπό να αντικαταστήσουμε το σύνολο των σταθερών υπολογιστών, το σύνολο των desktop από, αυτούς, από αυτές τις υβριδικές συσκευές που θα μας επιτρέψουν να εργαζόμαστε σε ψηφιακό περιβάλλον εργασίας, να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, σε ένα ενιαίο περιβάλλον και άρα να μπορεί κανείς να κάνει την ίδια δουλειά τόσο εντός όσο εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες. Το κόστος αυτών των συσκευών ανέρχεται σε 1.400 ευρώ περίπου. Και ε, θέλουμε να εγκαταστήσουμε 9.000 300 τέτοιες συσκευές, ήδη έχουν κατασταθεί 2.000, οι βουλευτές έχουν, έχουν εξοπλιστεί και θέλουμε να ενισχύσουμε τον εξοπλισμό αυτό και να δώσουμε αυτή την υλικοτεχνική υποδομή και στους βοηθούς. Είναι ένα σχέδιο που εκτείνεται σε βάθος ε, χρόνου ετών Ξεκινήσαμε φέτος, το 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε συστηματική αντικατάσταση των desktop, των σταθερών υπολογιστών γραφείου κάθε χρονιά και προσδοκούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Δεν θα αντικαταστήσουμε ένα desktop, ένα υπολογιστή γραφείου από μία υβριδική συσκευή, αλλά πολλούς υπολογιστές γραφείου από μία υβριδική συσκευή, γιατί μέσα στη διοίκηση εργαζόμαστε σε ένα, δύο, τρει διαφορετικούς χώρους εργασίας και ε, οι βουλευτέ βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς χώρους εργασίας, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και κάθε φορά έχουν ε, μηχάνημα πάνω στο οποίο δουλεύουν, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τον αριθμό των συσκευών και αυτό θα μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση δεν θα αντικατασταθούν μόνο οι σταθεροί υπολογιστέ γραφείου από φορητού, αλλά θα μειωθεί και το κόστο διαχείριση όλου, αυτού του εξοπλισμού του υλικοτεχνικού. Έχουμε περίπου 18.000 υπολογιστέ που έχουν εγκατασταθεί ε, στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να μειώσουμε το τεράστιο όγκο εργασίας που συνεπάγεται η διαχείριση όλων αυτών των συσκευών ε, και για και να έχουν και οι βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού κινητές συσκευέ. Θα μειωθεί και ο αριθμός δηλαδή. Και αυτό σημαίνει εξοικονόμηση. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να δώσω το λόγο στον κύριο Έλιο Γκαρότσα από τη Γενική Διεύθυνση SAFE. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη DG Safe, τις μεθόδους και τα σημεία αναφοράς με βάση τα οποία λειτουργεί αυτή η Γενική Διεύθυνση που είναι η πιο νεοσυσταθήσα. βασικό τη μέλημα είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των ατόμων και των αγαθών εντό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μειώσει τους κινδύνου και να προσφέρει ένα περιβάλλον εργασία γαλήνιο, ήρεμο και ασφαλές για τους βουλευτές και το προσωπικό επιτρέποντας τη διοίκηση, στο θεσμικό όργανο να παραμείνει ανοιχτό ως κοινοβούλιο, να επιδεικνύει τη διαφάνεια που το χαρακτηρίζει. Η Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας, λοιπόν, έχει ένα συνολικό κόνσεπτ ασφάλειας, μια έννοια για την ασφάλεια την οποία έχει εγκρίνει το Προεδρείο και έχει επικυρώσει τη στρατηγική της. Αυτή η στρατηγική κινείται σε πέντε βασικούς πυλώνες. Εσωτερήκευση, επαγγελματισμός, νέες τεχνολογίες, αξιολόγηση κινδύνου και κουλτούρα ασφαλείας. Εσωτερήκευση σημαίνει ανάληψη υποχρέωσης για την, εσωτερική, για την ασφάλεια από ε, τη διοίκηση, από το εσωτερικό και όχι ανάθεση σε τρίτους. Γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και στον προϋπολογισμό προβλέπεται να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα και για το Λουξεμβούργο. Υπήρξε καθυστέρηση ε, με το Λουξεμβούργο μόνο και μόνο επειδή περιμέναμε τις εξελίξεις ε, με την πολιτική για το κτηριακό. Δηλαδή δεν κάναμε δράσεις ακόμα ασφάλειας γιατί εκκρεμούσε το θέμα του κτηριακού, το οποίο θα ολοκληρωθεί φέτος. Το Κοινοβούλιο διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή το επίπεδο του επαγγελματισμού μας συγκρίνεται με επάξια με το επίπεδο ασφαλείας στα εθνικά κοινοβούλια και είχαμε την ευκαιρία να το αξιολογήσουμε αυτό και να το συγκρίνουμε και να το επιβεβαιώσουμε. Έχουμε tailored security, δηλαδή ασφάλεια αναπερίπτωση με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Κάνουμε αξιολόγηση κινδύνου κάθε φορά και προβλέπουμε σχέδιο ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες. Έχουμε νέες τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασιζόμαστε με ένα σχέδιο δράσης πενταετίας 2015-2020, το ολοκληρώσαμε και και μπορούμε πλέον να βασιστούμε στις νέες τεχνολογίες και έχουμε προβλέψει τέτοιου είδου αίτημα στον προπολογισμό του 2021. Τώρα το νομικό πλαίσιο είναι απολύτω σαφέ. Δουλεύουμε με διαφάνεια. Το 2018 το Προεδρείο ενέκρινε τη νομική μα βάση και το νομικό μα πλαίσιο για να μπορεί η Γενική Διεύθυνση Ασφαλεία να λειτουργήσει, η DG Safe και ε, όλοι αυτοί οι κανονισμοί έχουν δημοσιευθεί και ανακοινωθεί δεόντω. Έχουμε τρεις γενικές διευθύνσεις, δύο λειτουργικές επιχειρησιακές, μία οριζόντια η αρχιτεκτονική δομή βασίζεται στις συνέργειες και στις συνεργασίες μεταξύ όλων των τμήματων και υπηρεσιών, ε, διότι έχουμε το εξής απόφθεγμα, μία είναι η ασφάλεια και δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί, είναι μία και Έχουμε προκλήσεις ατυπικές, πολύ διαφορετικές. 80% του προσωπικού είναι με συμβασιούχους, είναι προσωπικό που λειτουργεί 24 στο 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Άρα η αρχιτεκτονική δομή είναι κάπως διαφορετική αφού οι άλλες υπηρεσίε έχουν κυρίως μονίμους και όχι συμβασιούχους. Και για να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας, συνεργαζόμαστε διαθεσμικά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και έχουμε και πολύ σημαντική συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Κάποια νούμερα τα ακούσατε χθε από το Γενικό Γραμματέα. 10.000 άνθρωποι μπαίνουν στα κτίρια κάθε μέρα. Το 2019 είχαμε ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Το 2019 4.000 εκδηλώσεις οργανώθηκαν εντός των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 250.000 επισκέπτες ε, συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις και είχαμε και 700 ε, επίσημες επισκέψεις βάσει πρωτοκόλλου και ούτω καθεξής. Ο προϋπολογισμός μειώνεται και πέφτει, μειώνονται τα ποσά στην επιχειρησιακή γραμμή του προϋπολογισμού, όμως επειδή έχουμε αναλάβει εσωτερικά το θέμα της ασφάλειας και στο Λουξεμβούργο, αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τους συμβασιούχους και γι' αυτό ο προπολογισμό φέτο είναι ίδιο και δεν έχει ούτε αύξηση ούτε μείωση σε σχέση με πέρσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σαστέλ. Και εγώ σα ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή την εσωτερική ε, ανάληψη τη υποχρέωση για την ασφάλεια στο Λουξεμβούργο και για την πρόσληψη συμβασιούχων για τη λειτουργία τύπου 1. Και θέλω να σα θέσω το εξή αφελέ ερώτημα. Αντικειμενικά φαίνεται αφελέ και το παραδέχομαι ανακαλύπτουμε αυτή την εσωτερική ανάληψη της ασφάλειας μέσα από τον προπολογισμό του 2021. Όμως, η ειδοποίηση για τις κενές θέσεις δημοσιεύθηκε χωρίς να έχει συζητηθεί πουθενά στην αλυσίδα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό. Πώς το εξηγείτε. Το γεγονός ότι η ειδοποίηση για κενές θέσεις έχει δημοσιευθεί έχουν δημοσιευθεί πολλές φορές αυτά για πολλές θέσεις, ενώ είμαστε στην αρχή του εγχειρήματος αυτού για τον προϋπολογισμό. Πολύ καλή απόφαση. Μου επιθυμίζει να μου επιτρέπει να σας επιθύσω ότι την απόφαση αυτή την πήρε το Προεδρείο το 2012. Να αναλάβουμε δηλαδή εσωτερικά το θέμα της ασφάλειας και το πράξαμε ε, για το Στρασβούργο και για τις Βρυξέλλες. Και καθυστερήσαμε να το εφαρμόσουμε για το Λουξεμβούργο λόγω του ότι περιμέναμε τις αποφάσεις για το κτηριακό. Θέλαμε να ε, συνδυαστούμε και να συμπορευτούμε με αυτές τις εξελίξεις για τα κτηριακά. Η εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό είναι εμφανής, είναι ελαφριά, αλλά υπάρχει. Ένα εκατομμύριο ευρώ εξοικονομείται για το Λουξεμβούργο, συνολικά. Και αυτό είχε προβλεφθεί στο παρελθόν. Διατηρήσαμε την εξοικονόμηση. Δηλαδή το 2015 με 2020 φάνηκε ξεκάθαρα ότι το γεγονός ότι δεν αναθέτουμε την ασφάλεια σε τρίτους και την αναλαμβάνουμε εσωτερικά είχε θετική επίπτωση στον προϋπολογισμό Κάναμε εξοικονόμηση και για το Στρασβούργο και για τις Βρυξέλλες και το ίδιο ε, θα συμβεί και με το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα. Αν όχι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά του 7 γενικού Διευθυντέ για τις πληροφορίες Μα έδωσαν και τα ερωτήματα τα οποία απάντησαν. Σα ευχαριστώ πολύ. We, we take a five minute break and then we can... Θα διακόψουμε για 5 λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε με τη συνεδρία τη Επιτροπή σε προπολογισμό σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2021. Uh, Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, συνεδρίαση της ε, Επιτροπής προπολογισμών. Συνεχίζουμε με την ε, μερίσια διάταξή μας στο σημείο 14, δηλαδή τις κατευθυντήρες γραμμές για τον προπολογισμό του 2021, τμήμα 3. Ε, αυτή λοιπόν η έκθεση είναι ένα σημαντικό έγγραφο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκφράζει την άποψή του σε ό,τι αφορά τον ε, επόμενο προπολογισμό, προκειμένου να ληφθεί εν λόγω άποψη υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία τη ε, πρόταση προπολογισμού. Διαφορετικά από ότι τα προηγούμενα έτη, οι διάφορε επιμέρου κοινοβουλευτικέ επιτροπέ θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του προκειμένου να προετοιμάσουν τι ονομοδοτήσει του σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση, προκειμένου ακριβώ να έχουμε, να μιλήσουμε, αν θέλετε, με μια ενιαία μια φωνή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δίνω τώρα ε, το λόγο στον κύριο Λάου Τουρού για να μας ε, παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σα παρουσιάζω το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ε, για τον προϋπολογισμό του 2021. Είναι κάπω ιδιαίτερο το έτος αυτό. Είναι το πρώτο έτος του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και είμαστε σε πλήρε διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, ε, εύχομαι η δουλειά μου να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους διαπραγματευτές για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρου, Όπως είπατε, οι κατευθυντήρες γραμμές είναι πολύ σημαντικός γιατί αποτελούν την έκφραση του Κοινοβουλίου και καταργήσαμε την εντολή για τον τριμερή διάλογο του Ιουλίου. Έτσι λοιπόν θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για πολύπλοκες διαπραγματεύσει, γιατί είμαστε σε οριστία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο Είμαστε στο τελευταίο έτος του προηγούμενου του δημοσιονομικού πλαίσιου πέρσι. Φέτος είμαστε στην οριστία και θα είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Είδαμε την ε, πρόταση του Σαρμισελ ε, για αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε για ένα προπολογισμό που περιορίζεται στο 1,07 του ΕΠΕ. Δεν ε, είναι και πολύ ισχυρό αυτό ο προπολογισμό. Έτσι λοιπόν, οι κατευθυντήριε γραμμέ μα θέλουν να βοηθήσουν τι καθολικέ, τι συνολικέ διαπραγματεύσει. Για τον προπολογισμό του 20, πέντε πολιτικέ ομάδε είχαν ε, μία ενιαία φωνή και γι' αυτό ε, μπορέσαμε να κερδίσουμε 1,9 δισεκατομμύριο επιπλέον. Γιατί πέντε ομάδε εργάστηκαν μαζί και κατέθεσαν κοινέ τροπολογίε και ελπίζω ότι θα έχουμε πάλι πέντε ομάδες που θα προβληματιστούμε από κοινού και θα παρουσιάσουμε κάποιες κοινέ τροπολογίες, ε, γιατί αν δεν είμαστε ενωμένοι, πολύ δύσκολο θα ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να στραφώ και στη διαπραγματευτική ομάδα, να τους πω ότι είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε. Ε, είναι πολύ ιδιαίτερη χρονιά φέτος, είναι το πρώτο έτος του νέου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, ε, μάλλον το 2021, όχι φέτος, με συγχωρείτε. Βλέπουμε ότι παρόλες τις φιλοδοξίες για μια πιο φιλόδοξη Ευρώπη, ε, η πρόταση του Σερμισελ ε, δείχνει παναχώρηση. Ταυτόχρονα θέλουμε να πετύχουμε σε δύο προτεραιότητες. Ε, θα εργαστούμε όλοι μαζί για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και η στόχοι είναι να πετύχουμε τον Green Deal και να έχουμε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%. 100 μέχρι το 2050. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει ε, να έχουμε θεσπίσει παντού, ε, παραδείγματο χάρη μέσα μαζική μεταφορά. Στι 14 Ιανουαρίου η ίδια η Κομισιόν ε, είπε ότι κάθε χρόνο λείπουν 34 έω 60 δισεκατομμύρια για να υλοποιηθεί το Green Deal και για τις προτεραιότητές μας. Ε, δεν ε, μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι όμως σκέφτονται ότι θα έχουμε νέο οικονομική κρίση αν δούμε το επίπεδο χρέου στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείες και το παγκόσμιο επίπεδο χρέου. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και ε, μας είπαν μάλιστα 32 οικονομολόγοι ότι δεν θα ξεφύγουμε από μια νέα οικονομική κρίση είτε φέτος είτε το 2021 και το του μας λέει ότι η επόμενη κρίση θα έχει 10 φορές χειρότερες κοινωνικές επιπτώσεις από την κρίση του 2008. Η κυρία Φόρντε Λάιεν ε, θέλει να θεσπίσει ένα σύστημα προστασίας ε, των ε, θέσεων εργασίας. Δύο φορές συνάντησα και τον κύριο Νικολά Σμίτ. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε αν επίκειται μια κρίση μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό να το έχουμε αυτό κατά νου προτεραιότητα δίπλα με τον Green Deal. Συγγνώμη, πολύ γρήγορα πήγα στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, οι ε, προτεραιότητε μα είναι να πετύχουμε την Πράσινη Συμφωνία. Στο έγγραφο τη 14η Ιανουαρίου τη Κομισιόν βλέπουμε με έκπληξη ότι η Κομισιόν έλεγε η ίδια ιδια τουλάχιστον λείπουν 500 δισεκατομμύρια και είχαμε και το θέμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Και εδώ βλέπουμε την πρόταση του Σερ Μισελ. Μας ε, είπε ότι πρόκειται για νέο χρήμα, ε, ότι πρόκειται για πρόσθετα κονδύλια, πέρα από αυτά που πρόσθεται η Κομισιόν. Ε, το, η Κομισιόν έλεγε χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και ένα η πρόταση που έρχεται από το Σερ Μισελ δεν έχουμε καν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια νέου χρήματο. Αν θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε το σταμείο τη Συνοχής, θα είναι δύσκολη η μάχη για να βρούμε αυτά τα νέα κονδύλια. Κατευθύνε γραμμή. Προτείνω να υπερασπίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι θέλουμε ένα περιπολογισμό που να ε, είναι ίσω με το 1,29 του ΕΠ, δηλαδή 192 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για το επόμενο έτος. Προτείνω να έχουμε προτεραιότητα για το κλίμα, το 30% του προπολογισμού να αφορά δράσεις για το κλίμα. Προτείνουμε επίσης να κάνουμε τα πάντα για να, πετύχουμε, να αποφύγουμε συγγνώμη, μια κρίση πληρωμών. Πριν 7 χρόνια είχαμε μια κρίση πληρωμών. Απριόριο έχουμε τώρα λιγότερους κινδύνους να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, έχουμε το σύστημα νησιν 1, νησιν 2, νησιν 3. Αυτό που ζητάμε 124 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για του χρόνου για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο. Και επίση η Κομισιόν ε, να μα ε, προτείνει ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη ε, και αν δεν ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει στο δημοσιονομικό πλαίσιο να μην μπλοκάρουν πληρωμέ. Άλλα δύο σημεία τώρα που θέλω να αναφέρω. Ξέρετε ότι έχουμε μία νέα ονοματολογία από επεξεργασία. Αυτή η ονοματολογία ενισχύει τη δυνατότητα να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο το Κοινοβούλιο και να μην έχουμε εντελώ αόριστου δείκτε που θα αποφασίζει η Κομισιόν ε, αντί για το Κοινοβούλιο και του πολίτε. Επιμένουμε λοιπόν αυτή η ονοματολογία να ενισχύσει το δημοκρατικό έλεγχο και για τι PPAs ε, τις πιλωτικές δράσεις και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχουμε σημαντικά πιλωτικά σχέδια στα οποία πρέπει να επενδύσουμε γιατί κάποια έτη ε, είχαμε κάποιες προτάσεις χωρίς ε, ιδιαίτερα επιχειρήματα και δυσκολευόμασταν να, διαλέξουμε μερικές ε, φορές κατατέθηκαν αυτά τα σχέδια χωρίς να γίνουν πραγματικές επενδύσεις. Και τελευταίο θέμα, το χρονοδιάγραμμα. Οι ε, τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 4 Μαρτίου. Νομίζω ότι θα έχουμε και μια συνεδρίαση για να εργαστούμε όλοι μαζί για τη βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται στις 30 Μαρτίου στο Στρασβούργο και η ψηφορία στην Ολομέλεια θα είναι στην δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος από του οικειώδει ε, συγκεκριτέ θέλει να πάρει το λόγο. Κύριος Ρέσλερ πρώτος λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στις απαρχές της δημοσιονομικής ε, διαδικασίας και θα είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία γιατί παράλληλα τρέχουν και οι διαπραγματεύσει ε, κατά τη διάρκεια όλου του έτου ε, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το πόσο σημαντικό είναι αυτό ο φάκελο. Αυτό εδώ ο προπολογισμό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε, ο τρόπο που θα μα επιτρέψει να μεταφράσουμε σε ε, πράξη όλες μας τις πολιτικές προτεραιότητες. Ευχαριστώ τον συγκητή για την προετοιμασία αυτού του σχεδίου χθες ό,τι αφορά τις βασικές μας πολιτικές προτεραιότητες. Από την ε, δική μα πλευρά, να σα πω ότι εγώ είμαι ο νέο αστιώτη συζητητή ε, για το ΕΛΚ, αλλά οι προτεραιότητε τη πολιτική μα ομάδα παραμένουν οι ίδιε. Δηλαδή, ε, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος χρειαζόμαστε έναν εξυγχρονισμένο προπολογισμό που να αντιποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Μία από αυτές και τις πιο επίγουσες είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι και η μόνη. Υπάρχει δηλαδή και ε, υπάρχουν και τεχνολογικές, ε, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, οπότε ε, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά θα πρέπει να επιμείνουμε στο να έχουμε έναν προπολογισμό ο οποίος θα είναι ε, σύγχρονος ε, και θα προσανατολίζεται προς το μέλλον, προς τις μελλοντικέ ε, γενιές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στο Εράσμου, φυσικά που αποτελεί από τι ναυαρχίδες αν θέλετε ως προς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από εκεί και μετά ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο προπολογισμό μας θα πρέπει να εκφράσει αλληλεγγύη, αλληλεγγύη σε διαφορετικά επίπεδα, καταρχήν σε επίπεδο Ένωσης που σημαίνει ταμεία συνοχής, κονδυλία συνοχής αλλά και σε διαγενειακό επίπεδο που με τη σειρά του περιλαμβάνει επενδύσεις σε πολιτικές ε, για την ε, νεολαία, πολιτικές απασχόλησης και οτιδήποτε έχει να κάνει με το Εράσμους, αλλά και όλες εκείνες οι δράσεις οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν στο να επιτύχουμε μια συνεκτική κοινωνία τόσο σε επίπεδο κρατών μενών, αλλά και αυτό είναι πιο σημαντικό, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, εγώ θα είμαι ε, ε, για τη σχετική γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής ε, ε και πρόκειται λοιπόν για με, συνήθως με από τις προτεραιότητες του ΕΛΓΑ πράγμα που θα παραμείνει και στο μέλλον έτσι σε ό,τι αφορά δηλαδή το σύντημα της μετανάστευσης για το οποίο χρειάζεται να υπάρξουν περαιτέρω επενδύσεις. Εάν λοιπόν υπάρχουν πολιτικές δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει τότε θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δεσμεύσεις όταν δηλαδή θα κληθούμε να κατανείμουμε τους περασμένους μας στο πλαίσιο του προπολογισμού. Αυτές λοιπόν είναι βασικές ε, κατευθύνσεις, αν θέλετε, οι ε, ε, βασικοί όροι στους οποίους θα βασιστούν οι προτάσεις τροπολογιών μας και βέβαια θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι πρώτες προτάσεις που θα γίνουν για τον προπολογισμό. Αναμένουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή όπως την είχαμε και πέρυσι. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τόρβαλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι μια ευχαριστη απέναντι στον συγητή για αυτό το σχέδιο έκθεσης που ε, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως προς το να ε, συμπεριλάβουμε τα κατάλληλα στοιχεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον προπολογισμό. Ε, και αυτό αναφέρεται και με τον κατάλληλο τρόπο, για παράδειγμα, μέσω και της αναφοράς του Green Deal. Ωστόσο, είμαι λίγο απογοητευμένος σε ό,τι αφορά αυτό το climate proofing μέσα στον τον προϋπολογισμό, δηλαδή ακριβώς ε, την λήψη υπόψη των συστηματών κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να περιλάβουμε ε, για παράδειγμα και άλλα στοιχεία, έρευνα και καινοτομία, Horizon Europe και υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως τώρα ανέφερε και ο εισηγητής έχουμε μια σειρά από μελλοντικέ προκλήσει που θα αντιμετωπίσουμε και πράγματι συμφωνώ ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και θα πρέπει κατά συνέπεια να αναφέρεται μέσα στι κατευθυντέ γραμμέ. Ωστόσο, αυτέ δεν είναι μόνε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Και νομίζω πω ε, είναι κάτι το, αυτό που θα πω, ε, κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι μα. Ε, δηλαδή, εάν δεν υπάρξει μια ανταγωνιστική βιομηχανία και μια ανταγωνιστική προσέγγιση που να συνοδεύσει το Green Deal, τότε το Green Deal δεν θα στεφτεί με επιτυχία. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εδώ να επιτύχουμε μια ισορροπία. Ναι, να ε, είμαστε αποφασιστικοί σε ό,τι αφορά την προώθηση του Green Deal, αλλά ταυτόχρονα να προσεγγίσουμε το Green Deal ε, με τρόπο ο οποίος θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να παραμείνει ανταγωνιστική, αλλά να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στο μέλλον. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω απευθύνεται περισσότερο στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και όχι στον ΕΣΥΔΕ, γιατί ε, το Συμβούλιο δείχνει να αντιμετωπίσει, αντιμετωπίζει δυσκολίες ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν ε, που θα πρέπει το να καταστήσουμε σαφές είναι ότι τα πράγματα δεν ε, παραμένουν ως έχουν. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ε, προπολογισμό που θα έχει υπερκοτοτηθεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να στεφθεί με επιτυχία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μας ε, και σε ό,τι αφορά και το Green Deal και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε μια, στο πλαίσιο μιας επικοδομητικής συνεργασίας με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους εστιώδεις εισηγητές ε, και αναμένω με ενδιαφέρον αυτή μας τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λαπούρτ. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, γενικοί προσωπικοί για τον προπολογισμό του 2021 δεν μας εκπλήσουν. Ίσως η έκπληξη είναι στο γεγονός ε, ότι αναφέρεστε σε μελλοντική κρίση οικονομική, αλλά αυτό όντως ε, λαμβάνεται υπάψη. Μιλάμε περίπου για το 1,3 ε, του ΕΠ. Αυτός είναι ο προπολογισμό που θέλετε σε αυτό το κείμενο για την περίοδο 2021-2027. Το Κοινοβούλιο ε, ζητά αύξηση προπολογισμού, όμως δύσκολο θα είναι να γίνει αποδεκτό αυτό από το Συμβούλιο. Και έχουμε και το Brexit, έχουμε κέρδη για 10 δισεκατομμύρια, όμως ε, δεν το βλέπω αυτό στο κείμενο. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από αυτό θα εξαρτηθεί ο προπολογισμό για το 2021. Θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή σας ε, στο εξή. Ε, στην αρχή το Κοινοβούλιο είχε μεγάλες διεκδικήσεις σε σημείο να αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ η συνθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας λέει ότι πρέπει να καθοριστεί ο προπολογισμό βάσει των προηγούμενων ετών. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, ο προπολογισμό του θα είναι ίδιος με το 2020 και αυτό θα είναι μεγάλη επαναχώρηση. Επίσης, είμαστε σκεπτικοί ε, στο αν μπορούμε να καλύψουμε τις προσδοκίες των πολιτών ε, και ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Μιλήσαμε για τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί για να βοηθήσουμε τους αγρότες να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό που ε, εντείνεται από τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Επίση, ε, θα πρέπει να δείξουμε ε, στου συμπατριώτε μα ότι δεν είναι οι μόνοι που κάνουν προσπάθειε, οπότε και εμεί πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Σκέφτομαι, παραδείγματο χάρη, το μηχανισμό με τη Ρερκία, το, τον προπολογισμό τη υπηρεσία εξωτερική δράση και άλλα. Έχουμε διάφορε δημοσιονομικέ θέσει που θα πρέπει να υποχωρήσουν τα επόμενα έτη. Για την προστασία του περιβάλλοντο, διάβασα ότι χρειάζονται περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο για να μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά τα αέρια του θερμοκηπίου ένα οικονομικό μοντέλο αποτελείται στο να ε, πουλάμε ένα προϊόν 10.000 ε, χιλιόμετρα μακριά. Αυτό αποτελεί οικολογική καταστροφή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Νομίζω ότι μας παρουσιάζει τις προκλήσεις και όπως είπε η συγητής είναι πολύπλοκο γιατί εργαζόμαστε σε έναν πρώτο προπολογισμό για το 2021 ο οποίος θα καθοριστεί από τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα για το πολιτιστικό οικονομικο πλαίσιο. Εγώ συμφωνώ με το γεγονό ε, να βάλουμε ως προτεραιότητα το θέμα τη στήριξης τη πράσινη συμφωνία, γιατί δεν είναι δυνατό ταυτόχρονα να λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο κύκλο και έχουμε νέε φιλοδοξίε με την Πράσινη Συμφωνία και να ξεκινάμε με βάση ένα προπολογισμό που θα αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχιση των όσων είχαμε μέχρι τώρα, ε, γιατί ή το θα έχουμε ό,τι κάνουμε συνήθω business as usual ή θα υπάρχει μια ρήξη. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήθελε μια ρηξη αυτο που καταλαβαινω ειναι οτι η προεδρο τη ευρωπαικη επιτροπη ηθελε μια ρηξη και το Κοινοβούλιο θέλει μια ρήξη και ε, οι διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σε διάφορες επικράτειες λένε επίσης ότι θέλουν μια ρήξη σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Έτσι λοιπόν, ε, ένας από τους πυλώνες του Green Deal είναι οι επενδύσεις. Να επενδύσουμε. Αυτό είναι πολύ καλό για την οικονομία, αλλά για να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή είναι η πρόκληση στο διακύβευμα. Δεν θα πρέπει όμως ε, να αντιτάσσουμε μια ε, φιλοδοξία οικολογική της Πράσινης Συμφωνίας ε, με αυτό που αποκαλούμε ανταγωνιστικότητα εδώ και 40 χρόνια. Αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους για την ανταγωνιστικότητα τα τελευταία 30 χρόνια, τότε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτός ο προπολογισμό θα μας χρησιμεύσει για να αναθεωρήσουμε την έννοια της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο. Δηλαδή μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να επιμείνουμε. Εγώ πιστεύω ότι επίσης είναι ενδιαφέρον να προλάβουμε τον κίνδυνο μιας μελλοντικής οικονομικής κρίσης. Τη τελευταία φορά όταν ξέσπασε ε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και δεν αδράξαμε την ευκαιρία ε, που είχαμε να αλλάξουμε μοντέλο. Τώρα είναι καλή ιδέα να προκαταλάβουμε τα πράγματα έτσι ώστε τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει κατά την άποψή μου πως να είναι στην προηγούμενη κρίση να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθά αυτή τη φορά. Και ένα τελευταίο σημείο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί πρέπει να προβλέψουμε ότι μπορεί να υπάρχει μπλοκή στις συζητήσει του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Πολλές ε, φορές ε, ε, εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να έχουμε ένα συνεκτικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όμως μπορεί να μην κατορθώσουμε να πεμπλοκάρουμε την κατάσταση. Πρέπει ουσιαστικά να πούμε ότι εμείς, το Κοινοβούλιο, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταιγίδα αν το Συμβούλιο δεν ακούσει τα δικά μας επιχειρήματα. Και τελικά από αυτό όμως να μην βλάψουμε μια σειρά δικαιούχους. Εγώ υποστηρίζω λοιπόν αυτό το πρώτο σχέδιο προπολογισμού και ευχαριστώ εκ νέου τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριο Τσάντσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Πράγματι, μιλήσατε για όλα τα ζητήματα κλειδιά που μας ενδιαφέρουν. Η δική μου πολιτική ομάδα, το ECR, θα υποστηρίξει το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά αυτές τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Πράγματι, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι σημαντικός στις διαπραγματεύσεις, γιατί το διακύβευμα είναι ο προπολογισμό για την επόμενη επταετία. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι υπάρχει διχογνωμία στην Ευρώπη. Υπάρχουν τα παλιά κρατημέλη, υπάρχουν τα νέα κρατημέλη. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει να καλυφθούν μεγάλα κενά σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, παραδείγματο χάρη στα μετακομμουνιστικά κράτη που μπήκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα για τη νέα πράσινη συμφωνία, τον Green Deal. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε και αυτό το θέμα, όμως εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν αδυναμίες εδώ, γιατί μέχρι τώρα πολλά λόγια λέγονταν για τον Green Deal, όμως Νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την πραγματική υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Θέλουμε λοιπόν πολύ πιο συγκεκριμένε προτάσει εδώ. Και φυσικά εμείς θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις δράσεις ε, κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την αναγκαιότητα να μιλήσουμε για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι πολλά πράγματα έχουν ήδη γίνει και πολλές πρωτοβουλίες είναι υπό ανάπτυξη, όμως υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που μπορεί να ξεσπάσουν στο μέλλον. Η οικονομική κρίση που αναφέρθηκε προηγουμένω, μπορεί να έχουμε νέο μεταναστευτικό κύμα, παραδείγματο χάρη, που θα καταφτάσει στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα, μπο... θα θέσουν ίσω μεγάλα προβλήματα. Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευράπης. Κάποιες εβδομάδες πριν, εδώ στο Κοινοβούλιο, οι Αμερικανοί μας παρουσίασαν ε, τη νέα τους τεχνολογία για τα ενεργειακά συστήματα. Σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν λύσεις που ε, ουσιαστικά προσεγγίζουν τη λειτουργία ε, των μονάδων άνθρακα, αλλά χωρίς ε, εκπομπές. Τέτοιες τεχνολογίες λοιπόν είναι ένα και πιο διαθέσιμες. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας για να μην χάσουμε αυτή τη μάχη για την ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να χάσουμε τη δική μας θέση που είναι πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και νομίζω ότι το μέσο της ενέργειας ακριβώς θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στο σύνολο της κλιματικής ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε λοιπόν τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτά τα ζητήματα και στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Εμείς εκπροσωπούμε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, γνωρίζουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά και στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλης. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαρουτηρίου, τον εισηγητή μας, γιατί κάνει αυτό που είναι αυτονόητο και πρέπει να είναι αυτονόητο για όλους μας και για όλες τις πολιτικές ομάδες. Υποστηρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επειδή ο προϋπολογισμός του 2021 είναι η πρώτη χρονιά του νέου πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, έχει τεράστια σημασία να μην αρχίσουν από τώρα διάφορες πολιτικές ομάδες να παίρνουν αποστάσεις από αυτό που ψήφισαν. Σε δύο μέρες θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής. Και ο κύριος Μισελ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, παρουσίασε μια απαράδεκτη πρόταση για το νέο MFF, για το νέο πολιετή προϋπολογισμό, που σε ορισμένα σημεία είναι χειρότερη και από την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σασόλη, είπε καθαρά, εκφράζοντας τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, εμείς απορρίπτουμε την πρόταση του κυρίου Μισελ. Θα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Renew και το ECR τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ή θα αρχίσουμε από τώρα τις εκπτώσεις. Γιατί από αυτό θα κριθεί όχι μόνο ο προπολογισμός του 2021, αλλά η μάχη για το νέο MFF. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι έχει σημασία να δούμε και να αντιδράσουμε στην πρόταση του Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση του κυρίου Μισελ προβλέπει μεγαλύτερες μειώσεις και από την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας στην κοινή αγροτική πολιτική, κατά 5 δις μικρότερη, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, μείωση σε σχέση με τη Φιλανδική Προεδρία 300 εκατομμύρια ευρώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μείωση σε σχέση με την απαράδεκτη πρόταση Φιλανδικής Προεδρίας 650 εκατομμύρια ευρώ, στο πρόγραμμα Horizon Europe μείον 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, πιστεύω ότι οφείλουμε όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες, να στηρίξουμε τη βασική θέση του εισηγητή, που είναι προϋπολογισμός για το 2021 1,29 του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, δηλαδή 192 δις. Γιατί αν φύγουμε από αυτό και πάμε στη λογική των μεγάλων περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο, τότε δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ούτε το Green Deal, ούτε η κοινή αγροτική πολιτική, ούτε η περιφερειακή πολιτική, ούτε η καινοτομία και το Horizon, ούτε το Erasmus, ούτε όλα όσα ζητάμε ως Ευρωκοινοβούλιο γιατί ζητάνε οι πολίτες από εμά. Εμείς με αυτό το πνεύμα, το επικοδομητικό, θα στηρίξουμε την θέση του εισηγητή, θα καταθέσουμε τροπολογίες υποστηρικτικές και καλούμε όλες τις πολιτικές ομάδες να στηρίξουν αυτά που έχουν ψηφίσει στην Ολομέλεια. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη, και θα πρέπει και η Κομισιόν να πάψει να παίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Η Κομισιόν εμφάνισε μία πρόταση για της κυρίας Φόντερ Λάιεν για να χρηματοδοτηθεί απαιτούνται χρήματα και επομένως δεν είναι honest broker. Πρέπει να ζητήσουν και αυτοί, όπως ζητάει το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο να χρηματοδοτήσει αυτές τις πολιτικές. Γιατί αλλιώς κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you. Does the Commission want to add some comments to this? Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει να κάνει κάποια σχόλια από την πλευρά της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να χαιρετήσω αυτήν την ανταλλαγή απόψεων που λαμβάνει η χώρα σε ό,τι αφορά την δουλειά που ήδη έχει κάνει ο εισηγητή, σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήρε γραμμέ για τον προπολογισμό του 2021. Νομίζω πω τα ε, βασικά στοιχεία και οι βασικέ προτεραιότητε ήδη αναφέρθηκαν στο πλαίσιο τη συζήτηση που έγινε. Και ο στόχο ε, βέβαια εδώ τη επίτευξη του Ευρωπαϊκού Green Deal είναι ένα στόχο στον οποίο ασπάζονται όλοι με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα επιτύχουμε και τις ε, προποθέσει ε, προκειμένου να κινηθούμε προς την κλιματική ουδετερότητα, πράγμα βέβαια το οποίο με τη σειρά του έχει και συγκεκριμένες οικονομικές ε, συνέπειες. Και αυτό το σημείο και τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν θα ληφθούν υπόψη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τη προετοιμασία του σχεδίου προπολογισμού, τη πρόταση προπολογισμού και βέβαια θα συζητηθούν και περαιτέρω στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου που θα ξεκινήσει στα τέλη του Απριλίου προκειμένου ακριβώς να ε, ε τροφοδοτήσει αυτό το, το, το, κείμενο με τις ε, πολιτικές προτεραιότητες ε, του ε, Κοινοβουλίου τη συζήτηση για το σχέδιο προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα το επίπεδο της εκτέλεσης του προπολογισμού, και το να υπάρχουν δηλαδή τα απαραίτητα κονδύλια, ναι, εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια ε, και ε, φροντίζουμε ε, ό,τι έχει εγκριθεί στο επίπεδο του προπολογισμού να εκτελείται. Να απορροφούνται δηλαδή αυτά τα κονδύλια και βρισκόμαστε τώρα σε μια ομαλή κατάσταση και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε από την πλευρά μα ότι μέσα στο 2021 να υπάρξουν όλες οι ε, ε, πιστώσεις ε, πληρωμών που θα συναντεύσουν τις σχετικές εντράσεις. Αλλά βέβαια όλες οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στην στο σημερινό επίπεδο της εκτέλεσης του προπολισμού και στις προβλέψεις που μα έχουν διαβιβάσει τα κράτη-μέλη. Ε, Τέλο, να πω κάτι σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο εκτάξη ανάγκη, το contingency plan που έχει προταθεί. Εμεί θα κάνουμε αν μας ζητηθεί τη σχετική πρόταση, αλλά νομίζω πω θα πρέπει τώρα να εστιάσουμε όλε μα τι προσπάθειε στην επίτευξη μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε και ένα πολύ ε, σαφέ σημείο αναφορά και ε, προβλεψιμότητα για όλους τους ε, εμπλεκόμενου σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό. Και εδώ εμεί ακριβώ θα παίξουμε αυτόν τον ρόλο του honest broker, του αμερόληπτου αν θέλετε δηλαδή. Ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ε, προπολογισμού. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχολιά σας και τις συμβουλές σας. Ε, φυσικά θα τα λάβω υπόψη και θα τα συμπεριλάβω, όμως είναι περιορισμένο το πλαίσιο, δεν έχουμε πολύ χώρο και δεν υπάρχει μόνο το θέμα του κλίματος, ακόμη και είναι για την ανθρωπότητα. Έχουμε το θέμα των ΜΜΕ, του Εράσμου, της κοινοτομίας, αναφέρονται και όλα αυτά. Αλλά βέβαια το θέμα του κλίματος ε, είναι το πιο τεράστιο εργοτάξιο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ε, που συζητάμε για τέτοιες προκλήσεις. Ε, και έχουμε και ένα παρατηρητήριο στην Αμερική που εδώ και 60 χρόνια παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη του διοξιδίου του άνθρακα και σήμερα αν συγκρίνουμε τη δεκαετία του 60 αυξάνεται το διοξιδίου του άνθρακα τρεις φορές ε, ταχύτερα. Έτσι λοιπόν ε, βλέπετε ότι έχουμε και τις φωτιές στην Αυστραλία και πολλές άλλες συνέπειες και σε κάποια Μόνο κάποια χρόνια έχουμε στη διάθεσή μα και ήμουν και στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια τη διάσκεψης για το κλίμα και πραγματικά όλο ο κόσμο έχει στραμμένο το κλίμα στην Ευρώπη για να δει αν θα υλοποιήσει τον Green Deal ή απλώς πρόκειται για ωραία λόγια. Είπε η απλω προκειται για ωραια Δεφάνδελερ, θέλουμε να πάμε στο ε, φεγγάρι, παρέθεσε τον ε, Κέννεντι, Όμω ε, επί 15 θα πρέπει να ε, πολλαπλασιαστεί ο προπολογισμό ε, της ΝΑΣΑ για να τα καταφέρουμε αυτά. Ε, και νομίζω ότι αν πρόκειται να σώσουμε τον πλανήτη μας, αξίζει να έχουμε έναν υψηλό προπολογισμό όμως για να καθησυχάζω τον Κάρλο. Είχαμε βάλει φέτος όλα αυτά τα στοιχεία, συγγνώμη πέρσι όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί να μην τα βάλουμε και για του χρόνου. Υπάρχει και το θέμα της νεολαίας και της συνοχής. Όλα αυτά αναφέρονται, αλλά αν θέλετε να είναι πιο έντονα θα το κάνουμε. Η ερώτηση του Νίλση για το θέμα της έρευνας. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σου, αλλά το θέμα της έρευνας ήταν ένα από τα πιο σοκαριστικά θέματα, ε, που, γιατί η ομάδα του Σέρλ Μισελ έκανε σοκαριστική πρόταση και μας ε, είπε ότι ε, είχε βάλει 5 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος για πολύ ενδιαφέροντα ε, ουσιαστικά ε, προγράμματα και έργα και τελικά αντί για αυτό το ποσό έβαλε μόνο 250 εκατομμύρια. Είναι απαράδεκτη η πρόταση και δεν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του Green Deal και της ανταγωνιστικότητας. Νομίζω όλοι συμφωνούν 240 ε, δισεκατομμύρια σε πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση για πετρέλαιο και αέριο που έρχεται από ξένε χώρε. Αν καταναλώσουμε λιγότερο αέριο και πετρέλαιο και έχουμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα δαπανίσουμε λιγότερα χρήματα και αυτά τα χρήματα θα μείνουν στη δική μα επικράτεια. Είναι στοιχείο ανταγωνιστικότητα. Ε, έχουμε χωριά στα Πυρηναία, παραδείγματο χάρη, που χρησιμοποιούν τη βιομάζα αντί για αέριο για τη θέρμανση και αυτό δημιουργεί θέσει ε, κάθε νοικοκυριό πληρώνει λιγότερο ε, και δεν πάνε αυτά τα χρήματα στα ταμεία του Πούτιν. Ε, έτσι λοιπόν δεν ξεχνάμε την ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε ένα μοντέλο που να προστατεύει τον πλανήτη και την κοινωνική πρόοδο. Ήμουνα στην Κρενόμπλε και είπαμε ότι μονώσαμε ε, το κτίριό μου, έχω λιγότερο, μάλλον κρυώνω λιγότερο το χειμώνα και ζεσταίνομαι λιγότερο το καλοκαίρι και κερδίζω και χρήματα. Και το είπε αυτό ένας πολίτης, ε, όχι ένας ε, βουλευτής και σε όλα τα νοικοκυριά, στη Γαλλία, στην Πολωνία, στην Ιταλία. Αν πούμε στους πολίτες θα σας βοηθήσει η Ευρώπη για να μονώσετε την κατοικία σας ή την επιχείρησή σας, είναι προς ε, όφελος της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Ο Νίκολας ε, Σμι, το επίτροπό μας, μας είπε ότι η καταπολέμηση της φτώχειας ε, φυσικά συνδέεται και με την ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δράσουμε και υπέρ του κλίματος, υπέρ της ανταγωνιστικότητας και για την καταπολέμηση της ανέχειας. Ο Νικολά ήταν υπουργό στο Λουξεμβούργο και εργάστηκε για την ε, μηδενική μείωση της ενεργείας και εκεί πραγματικά εφαρμόστηκαν οι τρεις αυτές διαστάσεις. Τώρα για μετά το Brexit, ε, ήδη οι πόροι είναι το κύριο θέμα για να απαντήσω στην κυρία Λαπόρτ. Το θέμα του Brexit ε, εντάσσεται στις προβλέψεις και το Κοινοβούλιο έλεγε πάντα ότι το κύριο διακύβευμα αν θέλουμε ένα μεγαλύτερο προπολογισμό, είναι να πεμπλοκάρουμε του ίδιου πόρου. Αυτό είναι το θεμελιώδε ζήτημα. Μία φορά το μήνα πάω στο Βερολίνο, γιατί η Γερμανία θα είναι ηγέτη στι διαπραγματεύσει και ο επικεφαλή τη Μπουντουρδοκ είναι εντελώ εχθρικό σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάθε φορά λέει όχι σε μεγάλο προπολογισμό, αλλά έχουμε δύο εξαιρέσεις. Ε, λέει, ας κάνουμε τα πράγματα σωστά, ποια είναι τα προβλήματα που δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε σε κάθε χώρα και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ευρωπαϊκά και δεύτερον, προστασία του περιβάλλοντος, το κλίμα και προστασία των συνόρων. Και εκεί λέει ε, ότι θέλουμε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και με ίδιους πόρους και καθώς πιστεύω ότι δεν είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά αν πρόκειται για το κλίμα και για την κοινωνική δικαιοσύνη και αν μπορούμε να έχουμε ίδιους πόρους, μπορούμε να πεμπλοκάρουμε τις διαπραγματεύσεις. Ε, για το θέμα του κ. Κορμάν για την ερώτησή του αν μπορούμε να, να συνεχίσουμε το business as usual. Όχι, σίγουρα μας ε, ανησυχούν οι εξελίξεις σχετικά ε, με το διοξείδιο του άνθρακα και βλέπετε και εδώ και ένα γράφημα. Βλέπετε το συνολικό χρέος των ήπα από το 1950. Βλέπετε υπάρχει πρόβλημα, ε, υπάρχουν 2-3 εκατομμύρια, 600 δισεκατομμύρια παραπάνω χρέος. Και εδώ βλέπετε τι γίνεται στην Κίνα. Και σαν έναν σε αεροπλάνο που να, και οι δύο κινητήρες κάνουν θόρυβο. Δηλαδή είπα και η Κίνα που κινούν την παγκόσμια οικονομία. Το 2008 ξέσπασε η κρίση στην Αμερική, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα είχε φτάσει στην Ευρώπη. Και δεν μπορούμε να λέμε αφορούν αυτά μόνο την Κίνα ή τη ΣΥΠΑ. Και να αναφερθώ και σε μια ερώτηση που έχω για την Κομισιόν. Όταν ε, η κυρία Φαρντελέν και ο Σμιτ μα λένε ότι είναι προτεραιότητα να έχουμε ένα σύστημα ε, αντασφάλιση ε, για τι θέσει εργασία, μήπω η Κομισιόν θα μπορούσε να προχωρήσει εκεί. Μήπως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί όταν ξεσπάσει η κρίση όλα αυτά είναι εικονικά σήμερα και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Κύριε για την ισορροπία μεταξύ των διαφορών περιφερειών συμφωνούμε. Πολύ συχνά είχαμε τη συζήτηση αυτή. Δεν είναι μόνο το θέμα της Πολωνίας ή της Ρουμανίας. Σε όλες μας τις χώρες και στην Ισπανία έχουμε άδειε ε, περιοχές και περιοχές που αναπτύσσονται πάρα πολύ. Θα πρέπει ο προπλογισμός να τους ωφελεί όλους, είτε ζουν στην Ήπεθρο, είτε στην πόλη, είτε στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία θα πρέπει είτε το Green Deal ή οι πολιτικές καινοτομίας ή οι πολιτικές έρευνας να χρησιμοποιηθούν και οι ερευνητέ ε, έχουν ε, πολύ συχνά κέντρα εξαιρετικά και τα νέα κέντρα στην Πολωνία ή στη Ρουμανία ε, δύσκολα βρίσκουν χρηματοδότηση. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα και θα μπορέσουμε όμως να το λύσουμε αν έχουμε ένα προπολογισμό που θα βασίζεται στους ίδιους πόρους. Και πιστεύω επίσης ότι το θέμα του κλίματος είναι ένα θέμα που μας βρίσκει σύμφωνους ε, για προγράμματα ε, που μιλάμε ε, και εμεί οι Ισπανοί σοσιαλιστές και ο Πολωνός υπουργό του Κλίματος δεν συμφωνούν σε όλα, όμως συμφωνούν για τα προγράμματα που προτείνουμε για τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. στη Μόναχο ε, είχαν πει είναι κομματιασμένη η Ευρώπη, μεταξύ είπα και Κίνα. Υπάρχει όμω ο κίνδυνο ε, να ε, απεμπλοκαριστεί η κατάσταση στην Ευρώπη. Πρέπει να δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει καταλητικό ρόλο, ότι προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα που αλλάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούν θέσει εργασία. Και νομίζω ότι το κλίμα είναι ένα από του μοχλού για να δώσουμε νέα όθηση στην Ευρώπη. Για να κλείσω μετά όσο είπε ο κ. Παπαδημούλη. Όλοι συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή, είμαστε, ε, όμως είμαι πιο αισιόδοξο ε, από σένα. Πιστεύω ότι και οι πέντε ομάδες ε, καταδίκασαν την πρόταση του Μισελ και εργάστηκαν από κοινού οι πέντε ομάδες για ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Όπω και να έχει, ελπίζω ότι όλοι θα συνεργαστούμε. Μπορείτε να μου στείλετε τις τροπολογίες μέχρι τις 4 Μαρτίου και μετά θα έχουμε μια συλλογική συζήτηση για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας της Επιτροπής Προπολογισμών. Θέλω να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 2 Μαρτίου εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών.